We were waiting for you to turn up, Eugen. <laughs> Colleagues, as it's uh, nearly... Αγαπητοί συναδέλφοι, είναι σχεδόν 9 και 10. Ας αρχίσουμε. Πρώτον, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Θεωρώ ότι εγκρίθηκε. Λοιπόν, έχουμε ή μάλλον δεν έχουμε τις εξής γλώσσες. Βουλγαρικά, Δανέζικα, Εστονικά, Φινλανδικά, Ουγγρικά, Ιρλανδικά, Λετωνικά, Λιθανικά, ε, Μαλτέζικα, Πορτογαλικά, Ρωμανικά, Σλοβάικα και ε, ε, Σλοβενικά. Γιατί μόνο οι γλώσσες των τακτικών μελών έχουν προτεραιότητα. Λοιπόν, επίσης στο σημείο 4 η ενημέρωση για την ad hoc αντιπροσωπή μας στη Γεωργία θα αναβληθεί για μια επόμενη συνεδρίαση γιατί λείπει η πρόεδρός μας, η κυρία Φωτίγα. Λοιπόν, οπότε, εφόσον έχει κρυθεί η μέση διάταξη, περνάμε στο πρώτο θέμα στην μέση διάταξη. Πού είναι το σημείο 3, το πρώτο σημείο για συζήτηση. Η κινητικότητα των στρατιωτικών. Λοιπόν, έχουμε τους ομιλητές μας. Είναι ο Αγνού Μόλνα, που είναι πεπειραμένος έμπειρος για θέματα ε, αμυντικής πολιτικής στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης και ο Ζάλου Ικολσόν, που είναι βηματάρχης ε, στη DG Move. Ε, στις 28 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος παρουσίασαν το πρόγραμμα δράσης για την κινητικότητα των στρατιωτικών ένα πολύ θετικό βήμα για την αντιμετώπιση ενό ε, θέματο που είναι βασικό σημείο για την συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ και έχει να κάνει και, μερικά, και με μερικά από τα θέματα που συχνά συζητάει η Επιτροπή μας. Είναι και θέμα ε, ενός προγράμματος ΠΕΣΚΟ με επικεφαλή στην Ολλανδία και έχει αντιμετωπιστεί και στα πλαίσια των προγραμμάτων EDA για πολλά χρόνια και στα πλαίσια της ε, πρότασης της Επιτροπής για ένα νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρξει μια χρηματοδότηση 6 δισεκατομμυρίων προς αυτή την προσπάθεια. Για πολλά χρόνια οι στρατιωτικές πλευρές της ε, ε, υποδομής μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν παραμεληθεί και χαίρομαι που τώρα υπάρχει η προσπάθεια να διευκολύνουμε την ταχεία μετακίνηση των στρατευμάτων μέσω του κοινού δικτύου μεταφορών. Αυτό είναι ζωτική σημασία για τη συλλογική μα άμυνα και γίνεται ακόμη σημαντικότερο όσο προχωράνε τα γεγονότα. Θα παρακαλούσα του ομιλητέ μα να διευκρινίσουν πώ προτίθεται η Επιτροπή να ε, χρησιμοποιήσει αυτά τα προτινόμενα 6 δισεκατομμύρια. Είναι μεγάλο ποσό, θετική εξέλιξη, αλλά πολύ διαρωτώμεθα πώς θα δαπανηθεί. Οπότε, να δώσω το λόγο, πρώτα απ' όλα, στο συνάδελφο που είναι εδώ αριστερά μου, τον κύριο Μόλεναρ, που όπως σας είπα είναι ανώτερος εμπειρογνώμονας για θέματα αμυντικής πολιτικής στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δίνετε να παρουσιάσω αυτό το θέμα και ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι βεβαίω ε, ζωτική σημασία. Όπως είπατε, μετά την κοινή ανακοίνωση του περασμένου Νοεμβρίου που έθεσε το πλαίσιο για το πρόγραμμα δράση που ενεκρίθη τον ε, παρελθόντα Μάρτιο από την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπήρξε στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής με της Επιτροπής ε, της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και του Οργανισμού για την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Το πρόγραμμα δράσης θα διευκολύνει περισσότερο τις ε, ένοπλες δυνάμεις για να αντιδρούν ταχύτερα ανάλογα με τις ανάγκες μας και στα πλαίσια της κοινή πολιτικής ασφαλείας και άμυνας και διαφορών αποστολών και στα πλαίσια των εθνικών και πολυεθνικών δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, το, το πλαίσιο της ΕΝΤΑ αναπτύχθηκε από τους τρεις φορείς αυτούς και είναι αποτέλεσμα της δράσης της ε, ομάδας ad hoc ε, με εθνικούς εμπειρογνώμονες που εργάστηκαν στα πλαίσια του Οργανισμού Άμυνας στα τελευταία ε, χρόνια, του τελευταίους μήνε μάλλον, και με τη συνεργασία του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Τώρα θα πρέπει να εφαρμόσουμε πρώτα απ' όλα την πολιτική πλευρά, τι πολιτικέ προποθέσει που αυτή τη στιγμή εκπονούνται από το στρατιωτικό μας προσωπικό μαζί με τα κράτη-μέλη, την Επιτροπή και σε ε, διαβούλευση και με το ΝΑΤΟ όπου πρέπει. Η Στρατιωτική Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τις ε, στρατιωτικές προποθέσει που τον Ιούνιο του 2018 θα πρέπει να εγκριθούν από το Συμβούλιο και επίσης υπάρχει ανάγκη να γίνει διαβούλευση με τα ε, αρμόδια σώματα του Συμβουλίου για αυτό. Το πρόγραμμα δράσης μας θέτει ένα συνολικό πλαίσιο για τις ε, παρούσες και μελλοντικές δραστηριότητες της Ένωσης Πρωτοκρατών μελών με συγκεκριμένε προθεσμίες για να υπάρξει συνέπεια. Είναι άλλο ένα βήμα στρατηγικής σημασίας γιατί θέλουμε να υπάρχει στρατηγική κινητικότητα, γιατί είναι απρόβλεπτη η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια. Η Ένωση λοιπόν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κρατών μελών, δίνει βοήθεια μέσω των ε, διαθεσίμων ενωσιακών μέσων. Συνεργαζόμεθα βεβαίως και με το ΝΑΤΟ, που επίσης ε, ασχολείται ενεργά με τα θέματα αυτό. Η Επιτροπής, ε, στην Επιτροπή σας ακούσατε μια ενημέρωση γι' αυτό. Η δυνατότητα λοιπόν περισσότερης ταχύτερης κίνησης ε, των στρατιωτικών δυνάμεων είναι σημαντικό θέμα συντονισμού της Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Πρώτα απ' όλα λοιπόν πρέπει να συμμετέχουν όλες οι αρμόδιες ε, εθνικές ε, υπηρεσίες, υπουργεία κτλ. με σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας. Τελικά το κράτος αποφασίζει για την μετακίνηση των στρατευμάτων του. Πρέπει να υπάρχει συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών και της Ένωσης για παράδειγμα, στα πλαίσια της μόνιμης ε, δομημένης συνεργασία και να υπάρχει συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Και αυτό είναι βασική αρχή. Και όλες οι αρχές ε, της συνεργασία με τον ΝΑΤΟ ισχύουν. Θα ασχοληθούμε με τους εξιστομείς. Ο Ζωάν Λουί θα ενημερώσει περισσότερο υποδομές, θέματα διαδικαστικά και ρυθμιστικά, θέματα τελωνιακά, ΦΠΑ και ε, οι άδειε για διαμεθοριακή μετακίνηση. Υπάρχουν και μερικά άλλα νομικά θέματα και αντιμετώπιση των ε, κύβερνων απειλών. Είναι σημαντικό θέμα και αυτό σε αυτό το τομέα. Τα κράτη-μέλη πρέπει να συνεχίσουν να συμμετέχουν ενεργά. Είναι βασικό σημείο αυτό για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Για να μπορούν να μετακινούνται ταχύτατα οι ένοπλες ε, δυνάμεις. Η συνεργασία των κρατών μελών είναι σημαντική και αυτό γίνεται μέσω των αρμοδίων Υπουργείων και άλλων εθνικών αργών, αρχών. Η εφαρμογή του προγράμματος δράσης πρέπει να γίνει με ολιστικό τρόπο. Εξετάζουμε βεβαίως και τα προγράμματα του ΠΕΣΚΟ το πρόγραμμα του ΠΕΣΚΟ, του οποίου ηγείται η Ολλανδία, που σχετίζεται με τα κράτη-μέλη και τι παραπάνω πρέπει να κάνουν σε θέματα αρμοδιότητάς τους για να βελτιωθεί η δυνατότητα μετακίνησης των στρατιωτικών δυνάμεων. Βεβαίως πρέπει να εξακολουθήσει να εμπλέκεται και το ΝΑΤΟ σε αυτό το τομέα. Τέλος Ιουνίου έχουμε το, τη Σύνοδο Κορυφής ε, της Ένωσης, ενώ τον Ιούλιο έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ οι αρχές της αυτονομίας, ε, της λήψης αποφάσεων, της συμμετοχής όλων και του σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών μελών, φυσικά όλα αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Συνολικά λοιπόν, νομίζω ότι προχωράμε γρήγορα. Το πρόγραμμα δράσης ε, έχει καθορίσει τη διαδικασία για τα επόμενα χρόνια. Το ίδιο το πρόγραμμα δράσης είναι ένα βασικό θέμα το οποίο πρέπει να προχωρήσει πριν από τη συνάντηση κορυφής του ΝΑΤΟ Πρέπει όλα αυτά να εφαρμοστούν, να γίνουν πραγματικότητα με τη βοήθεια των κρατών μελών, του Κοινοβουλίου και όλων των εμπλεκομένων ενωσιακών αρχών. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν οι συνάδελφοι που βάλουν ερωτήσεις που σίγουρα έχουν και πριν υπησέλθουμε σε λεπτομέρειες, να δώσω το λόγο στον Ζαν Λικόλσον που όπως σας είπα είναι τμήματάρχης της μονάδας για τις υποδομές μεταφορικές στην Γενική Διεύθυνση ΜΟΥΒ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, αγαπη... αξιότιμα μέλη, το σχέδιο δράσης για τη στρατηγική κινητικότητα απορρέει από αυτό που στις περιστάσεις αφορά τη μεταφορά στατευμάτων και υλικού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι πολύ δύσκολο τώρα και αντιμετωπίζει πάρα πολλά εμπόδια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατασκεύασε την ενιαία αγορά, δημιούργησε μια αγορά, αλλά όσον αφορά τα θέματα στρατιωτική κινητικότητα, τα σύνορα εκεί σε αυτό το πεδίο υπάρχουν πάντα. Ποια ήταν η ιδέα του σχεδίου δράσεω, να χρησιμοποιήσουμε συνέργειε που μπορούν να υφίστανται μεταξύ πολιτικών τη Ενώσεω όσον αφορά πολιτικά ζητήματα από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά να δούμε ποιε είναι οι ανάγκε. ανάγκες και να παρουσιαστούν συγκεκριμένες ε, δράσεις που στηρίζονται επί πολιτικών ήδη καταρτισμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως παραδείγματι η πολιτική των μεταφορών. Αυτό το σχέδιο δράσεως εστιάζεται επί μικρού αριθμού δράσεων, όπου οι ευθύνες σαφώς καθορίζονται με ε, φιλόδοξες ε, προθεσμίες και στόχους. Στόχος είναι να υπάρξει μια συμβολή στην αμυντική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ο πρόεδρος Γιούνκερ άλλωστε το εξέφρασε αυτό στην ομιλία του όσον αφορά την κατάσταση της Ένωσης και θέλουμε να δώσουμε στους πολίτες ένα συγκεκριμένο παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ενώσης ε, που προστατεύει και αμήνεται. Κάποιες δράσεις προβλέπονται στο σχέδιο δράσης που άπτονται των διαφόρων πολιτικών της νόσους, άπτονται της πολιτικής μεταφορών, της πολιτικής των υποδομών από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά της πολιτικής μεταφορών των εμπορευμάτων, επικινδύνων εμπορευμάτων και επίσης άπτονται και άλλων πολιτικών ε, της Ένωσης. Η πολιτική των υποδομών στον πολιτικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εδράζεται επί των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, τα τέντη, ε, Όπως γνωρίζετε αυτές οι πολιτικές ε, διακρίνουν τρία επίπεδα. Ένα γενικό επίπεδο, το πλήρες, το comprehensive, που πρέπει να υλοποιηθεί μέχρι το 2050. Ένα κεντρικό δίκτυο, το core network όπως αποκαλείται, που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι το 2030 και νέα διαδρόμους. Αυτές οι πολιτικές στον πολιτικό τομέα συμπεριλαμβάνουν και τεχνικές παραμέτρους. Οι διάφορες υποδομές δηλαδή θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο πολιτικό πεδίο σε κάποιες παραμέτρους. Παραδείγματι το βάθος των καναλιών ή το μήκος των αποβαθρών. Σε θετικά θέματα προβλέπονται τρία στάδια από τη μία πλευρά πρέπει να καθοριστεί το αναγκαίο δίκτυο που είναι αναγκαίο για την στρατηγική κινητικότητα και διάφορες τεχνικές παράμετροι που είναι ε, αναγκαίες για την ε, στρατηγική κινητικότητα. Ο Αρνού ήδη αναφέρθηκε σε αυτό. Ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να καθοριστεί από το Συμβούλιο βάσει εργασιών του ΙΟΜΕΣ και αυτό θα πρέπει να γίνει να ολοκληρωθούν οι εργασίες μέχρι το καλοκαίρι καταρχήν. Βάσει αυτών των συνεταιρικών παραμέτρων και βάσει των δικτύων που θα καθορίζονται και αυτά επιστοτικής βάσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προβεί σε μια σύγκριση μεταξύ των δικτύων και των παραμέτρων και το δίκτυο των διευρωπαϊκών δικτύων, το TNT, και των παραμέτρων του TNT. Οι ε, διαφορές θα εντοπιστούν και αυτές οι διαφορές ε, θα ποσοτικοποιηθούν θα δούμε τι θα είναι αναγκαίο να υλοποιηθεί πέραν των δικτύων TENTI, ούτω ώστε να καλυφθούν οι στατιτικές ανάγκες σε τεχνικό επίπεδο και σε επίπεδο γεωγραφικών δικτύων. Αυτές οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα Χριστούγεννα τρέχοντος έτους. Τέλος, ένα τρίτο στάδιο θα εντοπίσουμε πιστούν οι υποδομές των δικτύων, οι υποδομές που θα είναι αναγκαίες για στρατιωτικούς σκοπούς, αλλά που μπορούν εξίσου να ε, έχουν και κάποιο συμφέρον υλοποιηθούν για πολιτικό στάδιο. Δηλαδή ε, θα μπορούμε να, μπορούν να χρησιμοποιούνται υποδομές για όλες τις χρήσεις. Έτσι ε, και εντάσσονται γέφυρες Φερρυπίν που πρέπει να στηριχθούν, υποστηριχθούν για στρατιωτικές ανάγκες αυτές οι γέφυρες αλλά αυτή η στήριξη επίσης θα είναι κάτι χρήσιμο και για τους πολίτες. Θα επιτρέπουν τη διέλευση φορτηγών που θα μπορούν να βελτιώσουν την, ε, τις μεταφορές και την κυκλοφορία στο πολιτικό επίπεδο. Σε χώρες όπου δεν αντιστοιχεί το εύρος και η ανοχή όπως είναι η Βυρική Χεσόνιστο, οι Βαλτικές χώρες, η Φιλανδία, να αλλάξουν τις διαστάσεις και τις αποστάσεις μεταξύ ε, των ε, ραγών των, ε, των τρένων για να μπορούν να, να υπάρχει διέρεση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο και σε πολιτικό επίπεδο στις μεταφορές σιδηροδρομικέ. Μπορούμε να έχουμε και πολυτροπικέ βάσεις που είναι αναγκαίε, σε αελημένε, αερολιμένες που θα είναι κάτι απαραίτητο και σε θετικό επίπεδο, αλλά και θα είναι κάτι χρησιμότατο και για την πολιτική των μεταφορών στον τομέα των πολιτικών. Αυτές οι υποδομές dual use, διπλής χρήσης θα εντοπιστούν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόβλεψε κυρία Πρόεδρε και αναφέρθηκε αυτό έναν προϋπολογισμό στις δημοσιονομικές προοπτικές, στις μελλοντικέ 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση των εν λόγω υποδομών που θα είναι αναγκαίες για στρατιωτικές ανάγκες αλλά και χρήσιμες υποδομές για τον πολιτικό τομέα. Αυτή η χρηματοδότηση θα υλοποιηθεί μέσω των κλασικών μέσων χρηματοδοτήσεως των υποδομών μεταφορών στον πολιτικό τομέα, το ΣΕΦ, το Connecting Europe Facility, θα χρησιμοποιηθεί, συναρτήσει των διαδικασιών που προβλέπονται από το εν λόγω μέσο. Πρόκειται περί πολιτικής εποφελούς για όλους, win-win, που θα επιτρέψει καλύτερη υλοποίηση των δικτύων για τον πολιτικό τομέα και πιο γρήγορα πολιτικά δίκτυα για των μεταφορών, σύμφωνα με το TNT και ζώμη του TNT και θα προσαρμοστούν αυτά τα πολιτικά δίκτυα στις στρατιωτικές ανάγκες. Ε, άλλες δράσεις προβλέπονται επίσης πιο μακροπρόθεσμες. Επί παραδείγματι, ή ε, ε, να προσεγγιστούν οι βάσεις δεδομένων μεταξύ του TNT tec της βάσης δεδομένων του ΤΕΝΤΗ και του ΝΑΤΟ. Και αργότερα να έχουμε κανονισμό για τα ΤΕΝΤΗ και στον κανονισμό, με την επικαιροποίηση του κανονισμού, να συμπεριλάβουμε και στόχους ε, των στατιωτικών μεταφορών. Ε, άλλος άξονας τώρα, δεύτερος, η μεταφορά εμπορευμάτων, επικινδύνων εμπορευμάτων. Τώρα τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετική νομοθεσία όσον αφορά τη μεταφορά στατιωτικών ε, προϊόντων από ότι τα επικίνδυνα προϊόντα. Ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως υπάρχει μια οδηγία. Η οδηγία αφορά τη μεταφορά επικινδύνων φορτίων, αλλά αυτή η οδηγία δεν ισχύει παρά μόνο για τις μεταφορές αυτών των ε, εμπορευμάτων του πολιτικού τομέα. Ποια είναι η ιδέα λοιπόν, και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνα θα το κάνει αυτό. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε μια απογραφή των διαφόρων κανόνων που υπάρχουν και ισχύουν σε επίπεδο εθνικό στον τομέα της μεταφοράς στρατιωτικών μεταφορών επικινδύνων φορτίων και μετά να δούμε κατά πόσο μπορούμε να βασιστούμε επί των κανόνων του πολιτικού τομέα, τι πρέπει να προσθεθεί σε αυτούς τους κανόνες του πολιτικού τομέα, ούτως ώστε και οι στετιωτικές μεταφορές επικινδύνων φορτίων να εναρμονιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν τα κράτη-μέλη αισθανθούν ότι υπάρχει ανάγκη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε επίσης να υποβάλει κάποια πρόταση νομοθετικού περιεχομένου, τόσο ώστε αυτοί οι κανόνες μεταφορών επικινδύνων εμπορευμάτων στον στρατικό τομέα ε, να καλυφθούν νομικά, όπως αρμόζει. Το σχέδιο δράσεως λοιπόν επίσης προβλέπει και κάποιες δράσεις που βασίζονται επί άλλων πολιτικών του πολιτικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, παραδείγματος χάρη, η πολιτική τελωνιακή. Είναι σημαντικό στον τομέα το στατιωτικό να διευκολυνθεί η προσωρινή εξαγωγή υλικού και η επανεισαγωγή αυτού του υλικού στη χώρα προελεύσεως. Ε, για την ώρα δεν υπάρχει τέτοιος κανόνας, δεν υπάρχουν τέτοιοι κανόνες στο στρατιωτικό τομέα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να διευκολύνει αυτά τα εγχειρήματα χρησιμοποιώντας το βαθμό του δυνατού ένα έντυπο που προέρχεται από το ΝΑΤΟ, το 302 όπως αποκαλείται, και να αναπτυχθεί ένα ειδικό έντυπο την υπόθεση που το 302, το έντυπο 302 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αυτό θα απαιτήσει πιθανότατα τροποποίηση της δευτερογενούς νομοθεσίας σε θέματα τελωνιακά και τη δημοσίευση και έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατευθυντηρίων γραμμών. Αυτό προβλέπεται σε πρώτο στάδιο να γίνει μέχρι το τέλος ε, τρέχοντος έτους. Άλλη πολιτική, η πολιτική στον τομέα του ΦΠΑ, επί του παρόντος η πολιτική, το καταβάλλεται το ΦΠΑ όσον αφορά τις αγορές σε περίπτωση θετικών επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ενώ εξαιρείται στα πλαίσια στατιωτικών επιχειρήσεων, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Ποια είναι η ιδέα λοιπόν ενδεχομένως να επεκταθεί αυτή η εξαίρεση που υφίσταται στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στις επιχειρήσεις στρατιωτικές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Άμυνας, της κοινή Ευρωπαϊκής Άμυνας. Τέλος, προβλέπεται κάποια δράση στο πλαίσιο της αδειοδοτήσεως, διελεύσεως συνόρων από στατιωτικούς φορείς, Cross-Border Movement Permission όπως αποκαλείται, που συμπεριλαμβάνει ε, τη διπλωματική άδεια, diplomatic clearance, απλούστευση σε επίπεδο εθνικό, να υπάρξουν, να δημιουργηθούν σημεία επαφής των αρμοδίων υπουργείων σε εθνικό επίπεδο και να τεθούν μέγιστες προθεσμίες για τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο εθνικό. Ε, εκεί και αυτός είναι ένας τομέας ο οποίος θεωρείται σημαντικότατος όσον αφορά τη στατιωτική κινητικότητα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Thank you very... Ευχαριστούμε και τους δύο σας. Ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις, ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες που ακούσαμε για τα σχέδια αυτά. Φαντάζομαι ότι οι συναδέλφοι θα έχουν διάφορες ερωτήσεις. Θα δώσω καταρχήν το λόγο στον κύριο Γκάλερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πολύ καλή πρωτοβουλία αυτή. Όντως μας ενδιαφέρει να μπορούν οι ένοπλες δυνάμεις να μετακινούνται ούτως ώστε να υπάρχει αξιοπιστή άμυνα. Εάν δεν υπάρχει επαρκή κινητικότητα των, στρατιωτικών δυνάμεων, τότε θα αποτύχουμε πριν καν ε, αναλάβουμε δράση. Οπότε, ρωτάω, έχω την εντύπωση ότι πριν από την ε, πτώση του τείχους, ε, το ΝΑΤΟ είχε τη δυνατότητα να μετακινείται πολύ πιο σύντομα. Σωστή αυτή η εντύπωση ή όχι. Μπορούσαμε να φτάσουμε στην πρώτη γραμμή άμυνας ε, μέσω της Γερμανίας Βεβαίως τώρα πρέπει να μετακινηθούμε πολύ μακρύτερα, πρέπει να μετακινηθούμε χιλιάδες ε, χιλιόμετρα, άρα και γεωγραφικά είναι πιο δύσκολο. Αλλά εσείς μιλήσατε για ΦΠΑ, για διπλωματική παροχή αδειών, μήπως στο παρελθόν ε, ήταν καλύτερες οι λύσεις που είχαν επιλεγεί, δεν θα πρέπει λοιπόν να βασιστούμε σε αυτές. Υπάρχει, μας είπατε, ένα έντυπο του ΝΑΤΟ, το οποίο θα αντιγράψουμε απλώς. Μα τι θα γίνει με τις ε, ουδέτερες χώρες. Για παράδειγμα, αν θέλει να πάει κανείς από την Τσεχία στην Ουγγαρία, είναι καλύτερο να περάσει από την Αυστρία και όχι να πάει μέσω Σλοβακίας. Δεν μπορούν να υπάρξουν συμφωνίες με τα κράτη που δεν συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ να υπάρχει, ξέρω εγώ, ένα έγγραφο για τη μετακίνηση στρατευμάτων που να το αποδέχονται και αυτοί. Επίσης, αναφερθήκατε στις γέφυρες και στη δυνατότητα ε, αντοχής που έχουν οι γέφυρες. Και εδώ υπήρχε στο ΝΑΤΟ παλιότερα πείρα. Μας λέτε ότι στα πλαίσια ενός ε, προγράμματος του ΠΕΣΚΟ θα μπορούσαμε να έχουμε τη σωστή σήμανση για τις γέφυρες μέχρι τα ανατολικά σύνορα της Ένωσης, που είναι βεβαίως ταυτόσιμα με τα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να θεωρήσουμε ότι αυτά τα σήματα για τη δυνατότητα αντοχής κάποιων υποδομών να ε, ε, υπάρξουν ενιαία γιατί υπάρχει μια επιδότηση 20% της Κομισιόν ή νομίζω για το ΠΕΣΚΟ 30%. Θα ήταν πολύ συγκεκριμένο αυτό. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Και άλλη μία. Γιατί από τη μία έχουμε τον εξοπλισμό και από την άλλη έχουμε ε, το προσωπικό. Ξέρετε, οι στρατιώτες μας είναι πολίτες της Ένωσης, απλώς κάνουν ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Δεν θα πρέπει να πούμε κάτι παραπάνω γι' αυτό, διότι δεν θέλουμε να αντιπαρατεθούμε οι μεν τους, δεν θέλουμε να συνεργαστούμε για την άμυνα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να γίνονται επικαλύψεις. Δηλαδή, ε, καλύτερα, δεν θα πρέπει να δυσχεραίνουμε την μετάβαση συνόρων που θα ήταν πολύ πιο απλή για τους απλούς πολίτες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λούσιν, η κυρία Λούσιν. Ευχαριστώ πολύ. Το είπε η Πρόεδρός μας. Θα υπάρξουν 6,5 δις για να βελτιωθεί λοιπόν η κινητικότητα των στρατευμάτων. Στον τελευταίο προϋπολογισμό μας, συγγνώμη, στις τελευταίες προοπτικές 14-20, προβλέπαμε 24 δις για υποδομές. Για την περίοδο 21-27 προβλέπονται μόνο 15, σχεδόν 15 δις. Και τώρα έχουμε και αυτά τα 6,5 για την ε, κινητικότητα των στρατευμάτων. Οπότε ρωτάω, αυτά τα 6,5 δις θα δαπανηθούν με βάση την ε, την, χρησιμότητά τους για τη μετακίνηση στρατιωτών δεν θα μπορούσε να υπάρχει διτή χρησιμότητα. Επίσης, βλέπουμε ότι η χρηματοδότηση άλλων προγραμμάτων θα περικοπεί για να χρηματοδοτήσουμε τώρα στρατιωτικά προγράμματα και βεβαίως αυτά τα 6,5 θα συμπληρωθούν και με τις, δαπάνε δαπάνες του ΠΕΣΚΟ. Το είπε και ο κύριος Γκάλερα. Αυτά είναι κυρίως για το ΝΑΤΟ δαπάνες. Και θέλουμε να έχουμε και ένα κέντρο στήριξης που θα δημιουργηθεί. Σωστά είναι όλα αυτά που λέω. Θα υπάρξουν τελικά περαιτέρω δαπάνε στα πλαίσια του προγράμματος ΠΕΣΚΟ. Τι επιπλέον ε, μέτρα θα χρηματοδοτηθούν και από πού θα προέλθουν αυτές οι δαπάνες. Για την ομάδα μου το σημαντικό θέμα είναι εάν πρόκειται κυρίως να αξιοποιηθούν κάποιες δαπάνες για στρατιωτικούς σκοπούς τότε θα πρέπει να δαπανηθούν με βάση αυτά που προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας. Ευχαριστώ. Κύριος Φρόιντς. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω τι να πω. Πρέπει να φέρω έντονες αντιρρήσεις στην ερώτηση που είχε θέσει ο κύριος ε, Γκάλαγκερ, ε, την οποία έθεσα εγώ γιατί αφορά τη δική μου χώρα και όχι τη δική σας, παλιά. Ε, σήμερα ε, φτάσαμε ήδη στο 2018 και όχι στο 38, δεν είμαστε στο 38 ακόμα. Να επαναλάβω την ερώτηση, υπό διαφορετική χρειά όμως. Μιλάμε για ένα καλό μηχανισμό για την στρατιωτική κινητικότητα. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, η αυστριακή ουδετερότητα όμως. Γι' αυτό λοιπόν ξαναθέτω το ερώτημα του Μιχαήλ κάπως διαφορετικά. Διερωτώ με. Έχετε ένα κάρο σχέδια στην Ευρώπη για τη στρατιωτική κινητικότητα. Το θέμα αυτό πόσο θα επηρεάσει τη στρατιωτική κινητικότητα. Οι Αυστριακοί έχουν συμμετάσχει σε αυτές τις συζητήσεις. Πώς τους πείσατε, αν τους πείσατε. Ή πώς θα μπορέσετε να τους πείσετε, αν δεν τους πείσατε, να συμμετάσχουν σε όλο αυτό το σύστημα και να, δημιουργήσουν, να μην δημιουργήσουν προσκόμματα. Ευχαριστώ. Και μια-δυο ερωτήσεις από πλευράς μου, μια και είμαι και πρόεδρος. Προς τον κύριο Μόνο. Καταρχάς, εσείς το θίξατε, αλλά δεν το σχολιάσατε επαρκώς. Μιλάω για τις υβριδικές απειλές. Θα ήθελα να μας δώσετε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για αυτές. Επίσης, μετά την ερώτηση του κυρίου Γκάλερ και του κυρίου Φρόντ και της κυρίας Λόζινγκ, για τα πολιτικά δίκτυα TNT. Θα υπάρξει μια διαφορά στην έμφαση. Ε, σε ό,τι αφορά τους, ε, τις οδούς ή τις γραμμές που έχουμε ήδη προβλέψει στα πλαίσια του TNT. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Θα απαντήσουμε τη σειρά. Α επανέλθουμε σε ερωτήσει του κύριου Γκάλερ. Να σας πω από πού ξεκινήσαμε και αν θα μπορούσαμε να είχαμε προβλέψει το πρόβλημα αυτό και να το είχαμε αντιμετωπίσει νωρίτερα. Η νέα έμφαση αυτή προέκυψε τα τελευταία χρόνια δεδομένη και τη έμφαση του ΝΑΤΟ στην αποτροπή και στην ε, συνειδητοποίηση ότι υπάρχει πρόβλημα στη μετακίνηση στρατευμάτων προσανατολά. Αλλά μην θεωρήσετε ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν κάναμε τίποτα. Ο Ευρωπαϊκός Αμυντικό Οργανισμός είχε διάφορα προγράμματα για να ενισχύσει μια συνεπτική προσέγγιση στην χορήγηση διπλωματικών αδειών. Είχε γίνει πολλή προσπάθεια ε, από τον οργανισμό αυτό επί χρόνια για να βρεθούν πιο αποτελεσματικοί τρόποι για το θέμα αυτό. Ε, και να αντιμετωπίσουμε όλες τις, ε, τις μεταφορές. Ε, να υπάρχει μια συστηματική προσέγγιση, ούτω ώστε να διευκολυθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Χερσαίες, εναέριες κτλ. Υπάρχει δουλειά λοιπόν που έχει κάνει ο Ευρωπαϊκός Αμυντικός Μηχανισμός, ε, Οργανισμός, συγγνώμη, αλλά υπάρχει μια νέα επιτάχυνση τα τελευταία χρόνια για τη θέση των ουδετερών, χωρών που καταλαβαίνω ότι σας απασχολεί, σας ανησυχεί να σας τονίσω ότι συνεργαζόμαστε με τον ΝΑΤΟ, αλλά τα 28 κράτη-μέλη αποφασίζουν στο Συμβούλιο και αυτά καθορίζουν τη δουλειά που θα κάνουμε και για τις στρατιωτικές ανάγκες. 28 συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων και η Αυστρία είναι μία από τις 28 χώρες. Είχαμε αρχικές συζητήσεις και μας παρουσίασαν τη θέση τους, οι Αυστριακοί. Όμως τόνισαν ότι δεν ε, ακολουθούν πούμε, το πλαίσιο του ΝΑΤΟ, έτσι προφανώς, και τις επιταγές του ΝΑΤΟ. Το άλλο θέμα είναι ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να διευκολύνουμε. Μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε και στους κανονισμούς και στις υποδομές και στις δια... διαδικασίες. Οι αποφάσεις τώρα για το αν θα δεχτούμε τα ξένα στρατεύματα να περνάνε μέσα από το έδαφος μας, ξένα θέματα προφανώς, έτσι. Αυτό είναι θέμα εθνικό τελικά, είναι εθνική απόφαση, δεν υπάρχει κανένας αυτοματισμός. Αν μια υποδομή χρηματοδοτείται μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων, δεν υπάρχει εμέσως, ας πούμε, η, η συνεννόηση, ας πούμε, ότι θα αφήσει τα ξένα στρατεύματα να πέρασουν μέσα από το έδαφο σου. Όχι. Όχι, δεν είναι αυτόματη αυτή η απόφαση. Ε, μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά σε κάθε περίπτωση θα αποφασίσουν οι αστυνομικέ αρχέ αν θα δώσουν το πράσινο φω ή όχι. Αποφασίζουν λοιπόν ένα περίπτωση. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν μια διάκριση. Προσπαθούμε να διευκολύνουμε, να προωθήσουμε υποδομές, ε, κανονισμούς που επιτρέπουν ε, την γρηγορότερη μετακίνηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση η απόφαση είναι εθνική ε, και αυτό, στο εθνικό επίπεδο αποφασίζουμε αν θα επιτρέψουμε ξένα οι δικά μας τα να μετακινηθούν. Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα της μόνιμης διαθρωμένης συνεργασίας, δεν θα πρέπει να μιλήσω εγώ για αυτή τη δουλειά, γιατί ηγείται αυτής της προσπάθειας η Ολλανδία και προεδρεύει στις συνεδριάσεις αυτές. Το θέμα είναι να δούμε τι μπορούν να συνεισφέρουν τα κράτη-μέλη ε, χάρη στις εθνικές ε, αρμοδιότητες ή γνώσεις ή πραγματογνωμοσύνη που έχουν, ας πούμε, για γέφυρες, για οτιδήποτε. Αλλά και διάφορα εθνικά θέματα, οι εθνικές αρμοδιότητες, ο κ. Γκάλερ παρεμβαίνει. Θα πρέπει να έχουμε εναρμονισμένα πρότυπα. Ε, δεν θα πρέπει όταν περνά στα σύνορα, ας πούμε, ε, να έχουμε τελείως διαφορετικά πρότυπα. Ε, σε επίπεδο ΝΑΤΟ δεν υπάρχουν καθόλου εθνικές αρμοδιότητες. Υπάρχει ομιμορφία. Αυτή ήταν η ερώτησή μου και για τα οικονομικά ήταν, υπήρχε μια σχετική ερώτηση. Κοιτάξτε, είναι το θέμα της συνοχής, είναι σφαιρικότερο θέμα μεταξύ Ευρωπαϊκή Ενώσεω και ΝΑΤΟ εθνικού επίπεδου και επίπεδου ευρωπαϊκού. Αυτό είναι στο επίκεντρο των προσπαθειών μας. Θέλουμε να υπάρξουν συνέργειες και να συνδεθούν οι διάφοροι τομεί εργειών. Για την ώρα έχει δρομολογηθεί το σχέδιο αυτό διαθρωμένη συνεργασία στο ειδικό τομέα τη ΠΕΣΚΟ από το Δεκέμβριο. Αναπτύσσονται ιδέες σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχουν προγράμματα που απαιτούν μεγάλη χρηματοδότηση. Οι ιδέες εξετάζονται για διευκόλυνση και επιτάχυνση διαδικασιών με έμφαση στις εθνικές αρμοδιότητες. Για ευρυδικές απειλές. Σημαντικό αυτό, πράγματι. Διαφορετικές οπτικές γωνίες απαιτούνται. Η στρατηγική κινητικότητα πρέπει να ενταχθεί στην προσπάθεια για τις υβριδικές απειλές. Αυτό το πλαίσιο εφαρμόζεται. Και εκεί εντάσσεται η στρατηγική κινητικότητα. Όσον αφορά ενδεχόμενα στα οποία είναι απαραίτητη η στρατηγική κινητικότητα σε περίπτωση κρίσεως, πιθανότατα θα έχει υβριδική μορφή αυτή η κρίση σε κάποιες περιστάσει η λήψη αποφάσεων δεν θα είναι τόσο σαφής, η κατανομή αρμοδιοτήτων δεν θα είναι τόσο σαφή. Σε αυτές τις περιστάσει όμως πρέπει κανείς να μπορεί να κινηθεί, να αντιδράσει. Αυτή είναι η ουσία τη σχέση με τις υβριδικέ απειλέ. Πού καταλήγουμε. Στην κατανομή, στην αντιμετώπιση σε επίπεδα. Στατηγικό επίπεδο, επιχειρησιακό επίπεδο, χρειαζόμαστε ασφαλή δίκτυα, χρειάζεται προστασία αυτών αν υπάρχει εφοδιοπομπή στρατιωτική που έχει κολλήσει στα σύνορα, διότι δεν προβλέπονται οι κατάλληλε διαδικασίε για να μετακινηθεί και να πάει στο επόμενο κράτο μέλο, τότε γίνεσαι ευάλωτο όσον αφορά τι υβριδικέ απειλέ. Οπότε χρειάζεται περισσότερη επεξεργασία το θέμα. Και αυτό θα γίνει στα πλαίσια τη κοινή ανακοινώσεω για τι υβριδικέ απειλέ. Αυτά. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να προσπαθήσω να εστιαστώ στο θέμα της χρηματοδότησης, αν μου επιτρέπετε, και να απαντήσω με ακρίβεια στις ερωτήσεις που τέθηκαν για το θέμα αυτό. Στις δημοσιονομικές προοπτικές, η πρόταση για αυτές έγινε από την Κομισιόν. Πριν από λίγες μέρες μόλις. Το ποσό που θα δοθεί στο ΣΕΦ, στην, στο χρηματοδοτικό μηχανισμό συνδέοντας την Ευρώπη, το κλασικό μηχανισμό, χωρίς να μιλήσουμε για στρατιωτικές ανάγκες, είναι 24,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν υπάρχει μείωση, λοιπόν, σε σχέση με τον προηγούμενο προϋπολογισμό. Αντίθετα, υπάρχει μια μικρή αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο προϋπολογισμό. 24,1 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το ποσό που υπήρχε και μέχρι τώρα. Επιπλέον, πέρα από αυτά τα 24,1 δις, υπάρχουν 6,5 δις που θα δοθούν για τις διπλής χρήσεως υποδομές, όπως λέγονται. Πρόκειται για υποδομές απαραίτητες για να υπάρξει στρατιωτική κινητικότητα, αλλά φυσικά θα χρησιμοποιηθούν και στο πολιτικό τομέα. Έχουν και τέτοια χρήση. Αυτά λοιπόν τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να, να χρηματοδοτήσουν υποδομές που θα είχαν αποκλειστικά στρατιωτικό χαρακτήρα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για να χρηματοδοτήσουν υποδομές στο δίκτυο TEN-T μη στρατιωτική φύσης, το κλασικό, που χρησιμοποιείται όμως και από το στρατό. Επομένω, πρόκειται πρόκειται για δίκτυα χρήσιμα και στον πολιτικό και στο στρατιωτικό τομέα. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά το ΣΕΦ, το χρηματοδοτικό μηχανισμό συνδέοντα στην Ευρώπη, να τον καταστήσουμε ένα μηχανισμό χρηματοδότηση των στρατιωτικών υποδομών. Αντιθέτω, ο μηχανισμό αυτό παραμένει βασικά ε, μηχανισμό χρηματοδότηση ε, πολιτικών υποδομών και το ποσό το οποίο πηγαίνει για τη χρηματοδότηση των υποδομών αυτών δεν αλλάζει. Επιπλέον, υπάρχουν τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ όμως που θα πάνε για τη χρηματοδότηση υποδομών που φυσικά θα έχουν ε, σημασία και στον πολιτικό τομέα και που θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν και από το στρατό. Επομένω, θα κερδίσουν όλοι. Με αυτά τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ, τα επιπλέον 6,5 εκατομμύρια, θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε περισσότερα και για τι πολιτικέ ανάγκε ε, στα πλαίσια των δικτύων TEN-T, των δικτύων μεταφορών, δηλαδή διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Παρότι αυτά τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ θα χρηματοδοτήσουν και υποδομέ που είναι απαραίτητε και για το στρατιωτικό τομέα. Ευχαριστώ. Έχουμε λίγο χρόνο που απομένει για το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης, οπότε έχετε ερωτήσεις ε, άλλες ε, συνάδελφοι. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι συνάδελφοι που δεν μίλησαν και που έχουν κάποια ερώτηση που θέλουν να υποβάλουν στους εμπειρογνωμονές μας. Ο Μάικλ. Με το θέμα κινητικότητας προσώπων, ατόμων όχι μόνο την κινητικότητα του υλικού. Ε, το θέμα της διπλωματικής αδειοδότησης. Υπάρχει προθυμία από πλευρά κρατών μελών να δεχτούν τους στατιώτες μας ως πολίτες τους που μετακινούνται για κοινό στόχο, κοινό σκοπό ή θεωρούνται παρήσακτοι, ξέρω πώς να το πω. ε, μάχη με μάχημες εχθρικές ε, μονάδες. Χρειαζόμαστε τις γραφειοκρατικές αυτές άδειες. Χρειαζόμαστε τα ονόματα των στρατιωτών των συνταγμάτων που μετακινούνται όταν λένε Henry, Hans ή Giacomo πρέπει να καταχωρηθούν οι στρατιώτες και αν ασθενήσει πρέπει να πάρει άδεια και αν μπει κάποιος άλλος θα πρέπει μέσω περίπλοκης διαδικασίας να προσθεθεί κάποιος στρατιώτης στον κατάλογο. Ποιος είναι ο στόχος σας. Τα κράτη-μέλη σας καθοδηγούν, αλλά μπορείτε να είστε και δημιουργικοί και να χρησιμοποιήσετε φάνταστες λύσεις για τη διευκόλυνση των κινήσεων. Δηλαδή να κινήσετε υπέρ της απλούστευσης των διαδικασιών και όχι να τις κάνετε πιο περίπλοκες. Λοιπόν, ο Τζέιμς και ο Johannes. Η κυρία Λούζινγκ έχει το λόγο. Ναι, μια συμπληρωματική ερώτηση. για το θέμα του προπολογισμού. Με συγχωρείτε, δεν ήμουν ποτέ καλή στα μαθηματικά. Ναι. Αλλά ίσως σας κατάλαβα λάθος. Ίσως όμως και όχι. Τώρα βλέπουμε ότι προβλέπονται 15 δις. Εσείς είπατε ότι θα έχουμε 24 δις. Δεν άκουσα καλά μήπως. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι συμπεριλαμβάνεται και τι εξαιρείται. Όντω όπως και στις προηγούμενες ε, προοπτικέ προβλέπονται 24 δις, συν αυτά τα 6,5. Είτε είναι μόνο 15 για μη στρατιωτικούς σκοπούς και επιπλέον 6,5 και αιτιολογούνται αυτά τα 6,5 γιατί είναι διπλής χρήσης. Πόσα ακριβώς προβλέπονται τώρα συμπεριλαμβανομένων ή εξαιρουμένων αυτών των 6,5 δις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, διευκρινιστικές ή απλώς ερωτήσεις, να θέσουμε στους εμπειρογνώμονές μας αυτές τις ερωτήσεις. Ή το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Γκάλερ, για την ερώτησή σας. Ένας από τους στόχους δεν είναι μετακίνηση εξοπλισμού και μόνο και επικινδύνων εμπορευμάτων αλλά και του προσωπικού. Μία από τις προτάσεις προς εξέταση είναι η συμφωνία για το καθεστώς των δυνάμεων καταστατικό των δυνάμεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι διαφορετική αντιμετώπιση των διωτικών από αυτή των πολιτών. Με το ΣΟΦΑΡΤ, με αυτή τη συμφωνία, αν κυρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη, όσον αφορά το καθεστώς των στρατιωτών μπορούν θετικέ δυνάμεις που είναι σαν ο μέλος να έχουν προστασία, να τυχάνουν προστασίας, να μπορούν να μετακινηθούν κλπ. Ε, απαντώ στην ερώτηση, να μπορούμε να μετακινούμε ε, δυνάμεις χωρίς να έχουμε μεγάλες δυσκολίες. Εσείς? Ναι. Η απάντηση είναι σαφέστατη. 24,1 δις προς χρήση αποκλειστικά για τον πολιτικό τομέα. Συν 6,5 δις για την χρήση dual use. Σύνολο 30,6 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το σύνολο. Σαφέστατο. Σαφέστατη απάντησή σας. Ευχαριστώ για τις πλήρεις και περιεκτικές απαντήσεις. Είπατε προηγουμένως κάτι και με οδηγεί στην ερώτησή μου. Στο σχέδιο δράσεως, τι συγκεκριμένες νομοθετικού περιεχομένου προτάσεις θεωρείτε ως αναγκαίες για τη διευκόλυνση της ε, στατιωτικής κινητικότητας. Απάντηση. Η πρόταση κανονισμού του Connecting Europe Facility θα λάβει υπόψη προφανώς το σχέδιο δράσης, το action plan και τη δυνατότητα χρηματοδοτήσεως ε, υποδομών διπλής χρήσεως θα υπάρξουν συγκεκριμένες διατάξεις ειδικέ του κανονισμού που θα αναφέρονται στο dual use. Εν συνεχεία, δεν υπάρχει απόφαση, εξαρτάται από τη βούληση των κρατών μελών συνεχιδοδοθεί. Στην περίπτωση επικινδύνων φορτίων φερρυπίν. Είναι δυνατόν πράξεις νομοθετικού περιεχομένου να θεσπιστεί αν τα κράτη-μέλη θεωρήσουν ότι υπάρχει με τέτοια ανάγκη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φρονεί ότι, φρονήσει ότι είναι κάτι χρήσιμο και κάποιος δεντρολογικός κώδικας ίσως ε, να είναι αναγκαίος και μια πρόταση ε, νομοθετικού περιεχομένου ότι αυτή η περίπτωση δεν θα είναι απαραίτητη. Το ίδιο για τον κανονισμό τι αυτό καθε αυτό μπορεί να θεωρηθεί χρήσιμο, να συμπεριληφθεί εντός των ε, παρουσών παραμέτρων κάποιες παράμετροι για τις υποδομές που είναι απαραίτητες στο δυτικό τομέα, το ώστε στο μέλλον νέες υποδομές οι οποίες θα κατασκευαστούν να λαμβάνουν υπόψη τις θετικές ανάγκες. Δεν αποκλείεται αυτό αλλά δεν είναι και βέβαιο βέβαια ότι ε, θα γίνει κάτι τέτοιο. Σίγουρα θα χρειαστεί η τροποποίηση της ε, δευτερογενούς νομοθεσίας όσον αφορά το θέμα του ΦΠΑ και των τελωνίων, αλλά όχι απαραίτητα η ε, πρωτογενής νομοθεσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Πρώτα απ' όλα που ήρθατε εδώ σήμερα το πρωί να μας μιλήσετε και να αποσαφηνίσετε τα συγκεκριμένα σημεία που καλύπτονται από τον τομέα της ειδικής κινητικότητας. Στα αρχικά μου σχόλια είπα ότι αυτό είναι ένα θέμα που εξετάζει σοβαρότατα η Επιτροπή μας και με ικανοποίηση βλέπει πρόοδο στον τομέα αυτό. Προσβλέπουμε στη συνέχιση του διαλόγου μας επί του θέματος. Σας ευχαριστώ εκ νέου. Συνάδελφοι, όσα ανακοινώθη προηγουμένως, το επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως αναβάλλεται η ενημέρωση για την αποστολή της ΕΝΤΕ στη Γεωργία. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι, διότι δεν έχουν καταφτάσει ομιλητές για το επόμενο σημείο που ακολουθεί μετά. για, το, για, τα στρατεύματα, για τους πολίτες που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις και την προστασία τους. Προτείνω ε, μια σύντομη διακοπή των εργασιών μέχρι τις 10.30 όπου θα είναι παρόντες όλοι οι ομιλητές για το συγκεκριμένο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Σας περιμένω να έρθετε στην ώρα σας και μισή ακριβώς για να ξαναρχίσουμε τις εργασίες μας. Ευχαριστώ.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

Yeah.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

Right, colleagues, as um, when we broke earlier with uh, Λοιπόν, συνάδελφοι, είχαμε διακόψει μετά τη συζήτηση του προηγουμένου θέματος και είπαμε ότι θα τα ξαναπούμε στις 10.30 για την ακρόαση για τα δικαιώματα των στρατιωτών στα κράτη-μέλη της Ένωσης. έχουμε υπερβεί το χρόνο που είχαμε πει. Πιστεύω ότι πρέπει να αρχίσουμε. Να αρχίσει λοιπόν η ακρόαση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ο Εμμανουέλ Ιάκομπς από το Euromill, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στρατιωτικών Ενώσεων είναι παρόν, θα μας κάνει μια παρουσίαση για τα δικαιώματα των στρατιωτών και επίσης ο William McDermott που είναι ο υπεύθυνος ε, του Κέντρου της Γενέβης για το Δημοκρατικό Έλεγχο των Στρατιωτικών ε, των Ενόπλων Δυνάμεων, συγγνώμη, Αυτή είναι η πρόθεσή μας να ενημερωθούμε για την κατάσταση των δικαιωμάτων. Όταν ε, πήγαμε στο Μαλί, τον Νίγηρα και τη Βοσνία και τη Γεωργία, διαπιστώνουμε ότι πολλοί άνδρες και γυναίκες ε, είναι μαζί στο ίδιο περιβάλλον, για τον ίδιο στόχο ως στρατιώτες, καταπολεμούν τον ίδιο εχθρό. Όμως δεν έχουν κατανάγει τα ίδια δικαιώματα για παράδειγμα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, οι υπηρεσίε που του παρέχονται και άλλες ανέσει που τους παρέχονται και ιδιαίτερα πώς ε, τους φροντίζουν όταν αποστρατευτούν για να ενταχθούν και πάλι στην κοινωνία τους. Θα μας πούν λοιπόν οι εμπειρογνώμονες για την ε, κατάσταση όπως έχει σήμερα και αν ε, σε ενωσιακό επίπεδο θα μπορούσαμε και θα έπρεπε να επιδιώξουμε κοινέ προδιαγραφές για τη φροντίδα για τους στρατιώτες όταν ε, είναι σε αποστολές από κοινού. Έχουμε πολλές απαιτήσει από τις ενοπλές δυνάμεις μας, θα πρέπει να διασφαλίσουμε και την, ε, το καθήκον φροντίδας όταν επιστρέφουν. Να δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Γιάκο και μετά θα ακούσουμε και τον κύριο Μαρτέρμο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ για την εισαγωγή σας. Σας ευχαριστώ που μας καλέσατε. Ευχαριστώ και τα μέλη της Υποεπιτροπής που μας καλέσατε για αυτή την ακρόαση. Νομίζω ότι είναι σημαντική αυτή η ακρόαση και είναι υποφελής για τους ε, στρατιώτες της Ευρώπης ή τους Ευρωπαίους στρατιώτες. Παρότι είναι ανήκουν σε εθνικούς του στρατούς, θέλω να τους λέω, να τους ονομάζω Ευρωπαίους στρατιώτες. Αλλά από τη στιγμή που πηγαίνουν σε αποστολές υπό την Ευρωπαϊκή Σημαία, θα ήθελα να τους αποκαλώ έτσι. Θα ήθελα εν συντομία να σας, παρουσιάσω τη EuroMIL, που είναι η Ευρωπαϊκή Οργάνωση ε, Στρατιωτικών Ενώσεων. Μιλάμε για ε, ενώσεις και συνδικάτα. Ε, θα επανέλθω σε αυτό. Ε, ιδρυθήκαμε το 1972. Τότε ε, στρατιωτικές ενώσεις όπως από τη Δανία, την Γερμανία και το Βέλγιο δημιουργήθηκαν. Και η Ιταλία μάλιστα συμμετείχε. Ε, περίεργο είναι αυτό γιατί ε, ακόμα και σήμερα ε, οι Ιταλοί στρατιώτες δεν έχουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε. Ε, αλλά ήδη από το 1972 ε, είχαν ξεκινήσει να εργάζονται και να δημιουργούν ε, οργανώσεις αυτή τη στιγμή ε, εκπροσωπούμε 34 ε, οργανώσεις σε 23 ευρωπαϊκές χώρες. Η EuroMill είναι μια οργάνωση που είναι εντελώ ανεξάρτητη. Αυτό σημαίνει ότι δεν εξαρτώμεθα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν εξαρτώμεθα από την Κομισιόν, ε, δεν έχουμε σχέση με σύνδεση άμεση με τον ΝΑΤΟ. Είμαστε μια οργάνωση που χρηματοδοτούμεθα από τις χρηματοδοτήσεις των μελών μας. Αυτό περιπλέκει λιγάκι τα πράγματα. να τα καταφέρνουμε. Ε, μπορούμε όμως να κάνουμε τη δουλειά μας και εκπροσωπούμε περίπου 500.000 ε, Ευρωπαίους στρατιώτες και τις οικογένειές τους. Αλλά γι' αυτό χρειαζόμαστε εταίρους, ε, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και η, ο, η ΟΑΣΕ, οι συνάδελφοι από την ΤΙΚΑΦ της Γενέβης, ε, με τους οποίους συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά και διάφορες άλλες οργανώσεις ε, και φορείς ε, στις Βρυξέλλες όπως το καγκουρού, ε, οι Ευρωπαίοι φίλοι, οι φίλοι της Ευρώπης κτλ. Επίσης, ε, έχουμε ένα συμμετοχικό καθεστώς στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στο ΟΗΕ, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή του ΟΗΕ, έχουμε ένα καθεστώς συμβουλευτικού χαρακτήρα. Ε, Προσωπούμε λοιπόν ενώσει και συνδικάτα στρατιωτών, ε, προωθώντα ε, τις, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα επαγγελματικά συμφέροντα των στρατιωτών. Οι αρχές που χρησιμοποιούμε στη δουλειά μας είναι η αρχή το, το ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πολίτε με ένστολη. Και αυτό δεν σημαίνει ότι ένα στρατιώτη τον θεωρούμε σαν να είναι ένα οποιοδήποτε άλλο πολίτη, έτσι, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσει. Θεωρούμε ότι είναι πολίτε που φοράνε μία στολή και κατά την άποψή μα έχουν όλα τα βασικά και θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίε όπω οποιοδήποτε άλλο πολίτη, ε, ο οποίο ασκεί ένα επάγγελμα. Δεχόμαστε βεβαίω ότι το στρατιωτικό προσωπικό κάνει μια ειδική δουλειά και μερικέ φορέ. ε, με ασκούν τα δικαιώματά τους, αλλά υπό περιορισμό. Αλλά υπό φυσιολογικέ συνθήκες θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικοί πολίτε όπως και οι υπόλοιποι από εμά. Επίσης, ε, το είπε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξάλλου, αυτό που λέμε κι εμείς. Τώρα, η κατάσταση στην Ευρώπη, ποια είναι. Αυτό που θεωρούμε ως ένα από τα βασικά στοιχεία είναι το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε, το δικαίωμα στην ε, έκφραση του προσωπικού των στρατιωτικών δυνάμεων, των στρατιωτών, δεν είναι η βασική συζήτηση μας σήμερα, έτσι, ε, αλλά στις ε, στρατιωτικές αποστολές η, για να πάει ένα στρατιώτης και να συμμετάσχει σε αυτή την αποστολή χρειάζεται προετοιμασία. στρατιωτικής φύσεως προετοιμασία, αλλά και προετοιμασία για τα δικαιώματά τους, για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας. Αυτό δεν μπορεί να το κάνεις μόνος σου, σαν άτομο. Όποιος, όπως οποιοδήποτε άλλος δημόσιος υπάλληλο ή οποιοδήποτε εργαζόμενος σε εργοστάσιο, σε εταιρεία, κανένας δεν μπορεί από μόνος του να προσπίζει αυτά τα δικαιώματα. Θα πρέπει κάποιος να σε εκπροσωπήσει. Κάποιοι άνθρωποι να εκπροσωπήσουν αυτούς τους ανθρώπους, τους στρατιώτε και να υπάρξουν συλλογικές συμφωνίες ε, και να βρεθούν οι καλύτερες ε, συνθήκες διαβίωσης και εργασίας για το καθεστώς ε, του προσωπικού αυτού. Υπό αυτή την έννοια θεωρούμε ότι έχουν το δικαίωμα ελευθερίας λόγου ε, και ελευθερίας του συνεταιρίζεστε. Φυσικά, θα δείτε ότι δεν ισχύει κάθε φορά παντού αυτό στην Ευρώπη. βλέπετε αυτό το χάρτη, βλέπετε διάφορες χώρες, ε, τις χώρες με κόκκινο, που δεν θα έλεγα ότι κρούν τον κόδωνα, <laughs> μας κρούν τον κόδωνα, αλλά ανησυχούμε λιγάκι, γιατί εκεί οι στρατιώτες, το προσωπικό γενικά δεν έχει αυτό το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε ε, ούτε σε στρατιωτική ένωση, ούτε σε συνδικάτα. Ε, μερικές φορές διαφοροποιούμε ανάμεσα στις στρατιωτικές ενώσεις και τα συνδικάτα. Ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά. Είναι ότι οι επαγγελματικές ενώσεις, οι ενώσει, μπορούν να εκπροσωπήσουν τους στρατιώτες ε, και θα πρέπει να είναι ο συνομιλητή των πολιτικών αρχών, ενώ ε, τα συνδικάτα είναι ε, μία ένωση που λειτουργεί συλλογικά για το συμφέρον των μελών της, ε, για τους ανθρώπους που εκπροσωπεί και κάνει πολιτικά δεσμευτικέ συμφωνίες με τις αρχές. Αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα ενώσεις και στα συνδικάτα. Σε ορισμένε από τις χώρες βλέπουμε ότι έχουμε συνδικάτα τα οποία ούτως ή άλλως δεν μπορούν να ασκήσουν αυτά τα δικαιώματα πλήρως, γιατί είναι συνδικάτα στρατιωτών. Και σε άλλες χώρες έχουμε στρατιωτικές ενώσεις ε, που λειτουργούν πολύ επαγγελματικά και λειτουργούν σαν να ήταν συνδικάτα. Εδώ αυτό που βλέπετε στο χάρτη είναι ότι σε διάφορες χώρες στην Ευρώπη οι στρατιώτες και το στρατιωτικό προσωπικό δεν έχουν αυτά τα δικαιώματα. Ε, στις χώρες με πράσινο έχουν δικαιώμα, συνδικαλιστικά δικαιώματα, ενώ στα, στις χώρες με κίτρινο έχουν το δικαίωμα να φτιάξουν ε, ενώσεις. Ε, σε ορισμένε χώρε αυτά τα δικαιώματα υπάρχουν εδώ και 100 χρόνια. Σε ορισμένε πολύ πρόσφατα. Στη Γαλλία, α πούμε, ε, μόλι το 2015 ε, πήραν ε, το δικαίωμα, απόκτησαν το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε. Όταν μία απόφαση το 2014 εναντίον της Γαλλίας μία και στην άλλη περίπτωση εναντίον, ήταν μια υπόθεση όπου συμμετείχε μία οργάνωση, αποφασίστηκε ότι η Γαλλία δεν μπορεί να αρνηθεί το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε Στου στρατιώτε. Δεύτερα, ε, επίσης υπήρξε και μια άλλη υπόθεση της Euromill εναντίον τη Ιρλανδίας ε, που αφορούσε την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Χάρτα και όπου η Επιτροπή για την Κοινωνική Χάρτα δήλωσε το Φεβρουάριο του 2018 ότι η Ιρλανδία δεν μπορεί να αρνηθεί τα δικαιώματα τα συνδικαλιστικά στους στρατιώτες. Είχαν το δικαίωμα να φτιάξουν ενώσεις εδώ και 20-25 χρόνια ε, και τώρα θέλουν να αποκτήσουν και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Ε, επομένως, αυτή η συζήτηση ε, είναι ανοιχτή σε διάφορα επίπεδα και ε, έχει γίνει δεκτό ότι υπάρχουν αυτά τα δικαιώματα για τους στρατιώτες. Το σημαντικό ποιο είναι, ότι όταν μιλάμε για τις συνθήκες εργασίας και τα, τα, τις κοινωνικές συνθήκες, πρέπει να υπάρχει κάποια εκπροσώπηση. Κάποιο πρέπει να κάνει εξ ονόματός τους αυτές τις συμφωνίες και έτσι συνδέουμε. Τα δικαίωμα, το δικαίωμα του συνεστερίζεστε και το δικαίωμα του να συμμετέχει σε συνδικάτο με τον κοινωνικό διάλογο. Γιατί μόνο όταν έχει το δικαίωμα να ενταχθεί σε μία... Το να έχεις μόνο το δικαίωμα να ενταχθεί σε μία ένωση από μόνο του δεν έχει νόημα. Μερικές φορές είσαι εκεί, ε, έχεις το δικαίωμα να ανήκεις, αλλά κάνεις να σε εκπροσωπεί. Θα πρέπει να συνδεθεί αυτό με τον κοινωνικό διάλογο, ε, διάλογος μεταξύ ισοτήμων. Αυτό σημαίνει σεβασμός ε, μεταξύ των ε, στρατιωτικών και πολιτικών αρχών, και των εκπροσώπων του, των στρατιωτών και του στρατιωτικού προσωπικού. Οι κοινωνικές και ε, συνθήκες και οι συνθήκες εργασίας ε, έχουν να κάνουν με τη χώρα προέλευσής τους, αλλά και τι γίνεται όταν ε, βρίσκονται σε αποστολές οι στρατιώτες αυτοί. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία είναι, στην περίπτωσή μας, για και μιλάμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι η εφαρμογή της ε, ενωσιακής νομοθεσίας ε, για τα κοινωνικά και εργασιακά θέματα στα κράτη-μέλη. Συχνά χρησιμοποιούμε το παράδειγμα της ε, ασφάλειας των κατοίκων και των συνθηκών εργασίας, όπου υπάρχουν προβλήματα εφαρμογής σε στρατιωτικό επίπεδο. Ε, για πολλά κράτη-μέλη. Κοιτάμε αυτές τις οδηγίες ε, και την ε, νομοθεσία, το στρατιωτικό προσωπικό. Βλέπουμε ότι δεν αποκλείεται από την οδηγία ας πούμε, για το χρόνο εργασία. Η οδηγία αυτή ε, αφορά την ασφάλεια και το χρόνο. Έτσι. Ε, βασικά οι δύο οδηγίες συνδέονται μεταξύ τους. Είναι περίεργο λοιπόν που έχουμε χώρες όπου μόνο η ασφάλεια και η υγεία ε, εφαρμόζεται, αλλά όχι ο χρόνο εργασία. Ε, όχι, θα πρέπει να εφαρμόζονται και δύο οδηγίε. Επίση η Κομισιόν πολύ πρόσφατα είπε σε μία ανακοίνωση ακόμα μια φορά, αλλά η οδηγία για το χρόνο εργασία θα πρέπει να εφαρμοστεί για το στρατιωτικό προσωπικό. Τώρα, το να συνδεθεί τι γίνεται ε, με μια αποστολή και μάλιστα αποστολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν στέλνουμε κόσμο ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε αποστολή. Ούτω ή άλλω αυτοί εντάσσονται και καλύπτονται από την εθνική του νομοθεσία οι άνθρωποι αυτοί. Αν τα κρατήματα δεν εφαρμόζουν, αρνούνται να εφαρμόσουν ή εφαρμόζουν μόνο μερικώ τα μέτρα για την ασφάλεια και την ε, υγεία, α πούμε, το χρόνο εργασία. Ε, αυτό σημαίνει ότι όταν βρίσκονται σε αποστολή οι στρατιώτε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν μαζί δουλεύουν υπό διαφορετικά καθεστώτα και εθνικέ νομοθεσίε. Ενώ υπάρχει μια ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα έπρεπε να του καλύπτει όλου. Αυτό είναι προβληματικό ήδη από μόνο του. Οι στρατιώτες καλύπτονται από την εθνική τους νομοθεσία. Και οι εθνικές νομοθεσίες πολύ συχνά ε, αρνούνται στους στρατιώτες διάφορα δικαιώματα μόνο και μόνο γιατί οι στρατιώτες δεν θεωρούνται ως ε, φυσιολογικοί εργαζόμενοι στη χώρα τους. Σε ε, επιχειρήσεις και αποστολές της ΚΠΑ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύουμε εμείς στη Euromil ότι θα πρέπει να έχουμε κοινά πρότυπα για το στρατιωτικό προσωπικό. Πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή άνθρωποι συμμετέχουν σε μια τέτοια αποστολή υπό την ε, Ευρωπαϊκή Σημαία, σε αποστολές της ΚΠΑ, τότε σε κάποια φάση θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου όλοι αυτοί οι άνθρωποι εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο, δουλεύουν υπό τις ίδιες συνθήκες. Σήμερα δεν ισχύει αυτό, όπως σας εξήγησα. Σήμερα καλύπτονται από τις εθνικές νομοθεσίες. Εμείς πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα πρέπει να έχουμε κοινά πρότυπα και να ξεκινήσουμε με τις ε, νοσιακές αποστολές, γιατί είναι το μόνο πράγμα που έχουμε σήμερα στα χέρια, που έχετε εσείς στα χέρια σας, και μπορούμε να ξεκινήσουμε με το να επηρεάσουμε σε Ευρωπα... από το ευρωπαϊκό επίπεδο το εθνικό επίπεδο. Αλλά και τα επόμενα χρόνια, αργότερα δηλαδή, θα μπορούσαμε μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να κάνουμε βήματα, ούτω ώστε οι στρατιώτες και το στρατιωτικό προσωπικό που αν που πηγαίνουν σε αποστολές της ΚΠΑ να δουλεύουν υπό τις ίδιες συνθήκες της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Δηλαδή. Τώρα, όλα αυτά μαζί, αν τα βάλουμε όλα αυτά μαζί, συχνά ακόμα την αντίδραση. Μα, ωραία, καλά είναι όλα αυτά, αλλά είναι δυνατόν ο, ο στρατός να λειτουργεί έτσι. Ο στρατός δεν υπάρχει εκεί για να πειθαρχεί και να υπηρετεί. Και αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση Φυσικά, εγώ επειδή είμαι στρατιωτικό και εκπροσωπώ στρατιωτικέ ενώσει, ε, δέχομαι ότι θα πρέπει να υπάρχει στρατιωτική πειθαρχία. Θα πρέπει να υπάρχει πίστη στι ε, ενοπλέ δυνάμει και σεβασμό ιεραρχία. Αλλά θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα σε αυτό και στο γεγονό ότι θέλουμε να εκπροσωπήσουμε τα συμφέροντα των μελών μα, που είναι στρατιωτικοί. Και θα πρέπει επίση εξ ονόματό του, θέλουμε επίση εξ να κάνουμε διαπραγματεύσει. Θα πρέπει να βρούμε την ε, σωστή ισορροπία. Και ε, πολλά παραδείγματα στην Ευρώπη που δείχνουν ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει. Είναι δυνατόν να βρεθεί αυτή η ισορροπία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπω σα είπα, έκανε διάφορα πράγματα στον τομέα αυτό. Ήδη στο παρελθόν, το 1984 ήδη, ε, το Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα για τα δικαιώματα των μελών των ενόπλων δυνάμεων και εν συνεχεία το 1995 ένα άλλο ψήφισμα για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και συνεχεία ένα ψήφισμα για την περίοδο 2004-2008 και είπαμε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν σταματούν στις πύλες ενός στρατοπέδου. Ε, και είναι, αυτό είναι η βασική αρχή που μας ε, ε κατευθύνει, ας πούμε, για τους έστωτους πολίτες. Ε, δεν σημαίνει ότι από τη στιγμή που μπαίνει στο στρατόπεδο πάβεις να είσαι πολίτες και κάποιος ο οποίος δεν έχει πια δικαιώματα. Αντίθετα, έχεις δικαιώματα. Επίσης, το πιο πρόσφατο ψήφισμα, και πολλοί από εσάς συμμετείχατε, ήταν το ψήφισμα ήταν για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση, όπου μας άρεσε πραγματικά το άρθρο 12 του ψηφίσματος, που ζητάει από τα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν το δικαίωμα του στρατιωτικού προσωπικού να δημιουργήσει επαγγελματικέ οργανώσεις ή συνδικάτα, ε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Αλλά και να τους ε, εντάξει σε ένα τακτικό κοινωνικό διάλογο με τις αρχές. Ε, σας είμαστε ευγνώμονες ε, ο, γιατί ψηφίσατε αυτό το ψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση και ευχαριστούμε κυρίως όσους υπερψήφισαν ε, αυτή τη συγκεκριμένη τροπολογία, αυτές τις τροπολογίες προς αυτήν την κατεύθυνση. Το μέλλον τώρα της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Έχω πει και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλοι αυτό έχουν πει και εδώ στο Κοινοβούλιο και σε διάφορες συνεδριάσεις ότι είναι ξεκάθαρο τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Άμυνα άλλαξε πολύ και ότι έγιναν πολλά για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, μάλλον ε, τα τελευταία 1,5-2 χρόνια, παρά τα προηγούμενα 15-20 χρόνια. Τα τελευταία αυτά χρόνια υπήρξε μια επιτάχυνση και πιστεύουμε ότι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία για να αποκτήσουν κοινωνικά δικαιώματα οι στρατιώτες και να υπάρξει συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό δεν σημαίνει πάρα αυτά ότι τα έθνη χάνουν την αρμοδιότητα που έχουν για τι αναπλές δυνάμει του. Να το πούμε ξεκάθαρα, γιατί αυτό μα το λένε και το ξαναλένε. Δεν σημαίνει ότι χάνουν την αρμοδιότητά του για το στρατιωτικό προσωπικό. Ε, απλώς θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο συντονισμό των συνθήκων ε, για το προσωπικό αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω αυτής της ιδέας για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση. Μέσω αυτού του πλαισίου. Ειλικρινά σας λέω, δεν ξέρουμε πού θα μας οδηγήσει η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση. Δεν ξέρω αν εσείς το ξέρετε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά ούτως ή άλλως το ψήφισμα υπάρχει και κάποιοι από εμά έχουμε ξεκάθαρες ιδέες για το μέλλον αυτό της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης. Ε, δεν συμφωνούμε όλοι φυσικά. Πάντως αλλάζουν τα πράγματα και αυτή η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση είναι επιτάπητος. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε επ' αυτής και θα προσπαθήσουμε, θα προσπαθήσουμε σε αυτό το πακέτο να βάλουμε και τις συνθήκες εργασίας και τις κοινωνικές συνθήκες για το στρατιωτικό προσωπικό. Ε, και αυτά να τα ρυθμίσουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν συνέχεια, η μόνιμη διαθρωμένη συνεργασία, η ΠΕΣΚΟ. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση χωρί να αναφέρουμε την ΠΕΣΚΟ. Α μην είμαστε αφελεί Όμω, Εμείς τουλάχιστον δεν είμαστε αφελείς και δεν πιστεύουμε ότι επειδή ξαφνικά υπήρξε η ΠΕΣΚΟ θα βρεθεί η μαγική λύση για όλα τα, τα προβλήματα τα επόμενα χρόνια. Αλλά είναι ένα τεράστιο βήμα αυτό. Αυτό που λείπει, κατά την άποψή μα, είναι ότι στη μόνιμη αυτή διαφορεμένη συνεργασία, τουλάχιστον σήμερα και στην αφετηρία της, δεν υπήρχε τίποτα για τα κοινωνικά δικαιώματα ή τα ανθρώπινα δικαιώματα των στρατιωτών. Φυσικά, έχουμε κάποια στοιχεία ε, του πρώτου πακέτου προγραμμάτων και τα δεύτερα, το, τη δεύτερη δέσμη θα την έχουμε ως ονούπο. Ήδη από το πρώτο πακέτο έχουμε κάποια, κάποιους προπομπούς που μιλάνε για κοινωνικά δικαιώματα κτλ. και για το συντονισμό των δικαιωμάτων ε, Υπάρχει ένα project για την ιατρική περίθαλψη, ας πούμε, που θα είναι πολύ σημαντικό, ειδικά σε κάτι επιχειρήσεις και τις αποστολές. Πώς θα μπορούσαμε δηλαδή να συνεχίσουμε να δεχόμαστε ότι όταν οι στρατιώτες μας πηγαίνουν όλοι μαζί διάφορα έθνη σε μια στρατιωτική αποστολή υπό την σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποια στιγμή, πάντα λέω το ίδιο παράδειγμα, έτσι, ελπίζω να μην συμβεί ποτέ, αλλά το λέω πάντως. Ε, είμαστε στην ίδια αποστολή για την Ευρωπαϊκή Ένωση με Ευρωπαίους στρατιώτες, με την Ευρωπαϊκή Σημαία στην στολή τους. Έχουν, ας πούμε, με ένα τζιπ ένα ατύχημα και έχουμε, ας πούμε, θεωρητικά έτσι, τέσσερις ανθρώπους τραυματισμένους με τον ίδιο τρόπο, που μπορεί και να πεθάνουν τελικά στην αποστολή αυτή. Πώς θα συνεχίσουμε να δεχόμαστε ότι αυτοί οι τέσσερις άνθρωποι ε, αντιμετωπίζονται τελείως διαφορετικά μόνο και μόνο γιατί καλύπτονται από την εθνική νομοθεσία του καθένας αυτό μπορεί να αφορά. Ε, μερικά κράτη, ας πούμε, μπορεί να τους ε, φροντίζουν πάρα πολύ αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους στρατιώτες και κάποιο άλλο κράτος μπορεί να μην κάνει τίποτα. Και μπορεί τελικά οι τραυματίες στρατιώτες να φύγουν από τις ενοπλές δυνάμεις χωρίς τίποτα στα χέρια τους. Ε, νομίζουμε ότι αυτό είναι το πιο επίγον θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει και εκεί τα προγράμματα της ΠΕΣΚΟ για την ε, ιατρική περίθαλψη ας πούμε, θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Τέλος και σημαντικό, τελευταίο και σημαντικό, ένα παλιό σημείο. Ήδη το 2009, το 2010, το Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχτηκε ένα ψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια ε, και την ΚΕΠΑ και εκεί είχαμε το SAFE. συγχρονισμένε ε, στρατιωτικέ δυνάμει Ευρώπη. Ε, μιλούσαμε για συντονισμό, για κοινέ ασκήσει και εκπαίδευση, για κοινωνικά δικαιώματα των στρατιωτών. Εμεί πιστεύουμε πραγματικά ότι αν βρούμε έναν τρόπο να συνδέσουμε τα προγράμματα της ΠΕΣΚΟ, τα οποία υπάρχουν επιτάπητο σήμερα και τα παλιά προγράμματα της, του ΣΕΙΦ, που δεν ε, υλοποιήθηκαν ποτέ στην πραγματικότητα, είναι από το 2009-2010 αυτά τα προγράμματα του SAFE. Αν προσπαθήσουμε να τα επαναφέρουμε. Ε, γιατί οι αρχές που υπήρχαν στο SAFE ε, συνδέονται με τα προγράμματα του ΠΕΣΚΟ και θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν για να γίνει καλύτερο συντονισμό στο μέλλον. Θέλω να κλείσω τώρα με την εξή ε, φράση. Το πιο σημαντικό που χρειαζόμαστε είναι μεγαλύτερο συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο κοινωνικά δικαιώματα και συνθήκες εργασίας πιο συντονισμένε για το στρατιωτικό προσωπικό. Και α ξεκινήσουμε με τις ε, ευρωπαϊκές αποστολέ. Είναι κατάλληλη στιγμή, είναι μια καλή λύση αυτή να δουλέψουμε σε αυτό το επίπεδο. Α, μιλάμε για στρατιώτε, οι οποίοι φεύγουν μαζί για κοινή αποστολή. Εάν έχουν το ίδιο καθεστώ από την αρχή τη προετοιμασία τη αποστολή μέχρι τη στιγμή που επιστρέφουν στη χώρα τους, αν τους δούμε ως Ευρωπαίους στρατιώτες και όχι εθνικούς στρατιώτες με εθνικά δικαιώματα, ε, θα έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα. Και εν συνεχεία σε μια δεύτερη φάση, ας πάμε ακόμα πιο πέρα και σε μια τρίτη φάση, ας πάμε ακόμα πιο πέρα για να συντονιστούμε ακόμα περισσότερο και εκτός ε, τέτοιου τύπου αποστολών. Αυτά, Πρόεδρε. Αυτά ήθελα να πω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βεβαίως είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Thank you, Mr. Jacob. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιάκομπ. Να καλωσορίσω και τους προσκεκλημένους μας και πολύ σύντομα θα σας παρουσιάσω, αλλά καταρχάς σας καλωσορίζω. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον, ε, στον William McDermott από την οργάνωση DICAF. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ όλους ε, που ε, είστε εδώ για τη συμμετοχή σας. Λέγομαι William McDermott. Η οργάνωση μου λέγεται DICAF. Βασίζεται στη Γενέβη, έχει έδρα τη Γενέβη. Τι είναι λοιπόν ο οργανισμός μου. Πριν ασχοληθώ με τα ανθρώπινα δικαιώματα του προσωπικού των όπλων δυνάμεων, η οργάνωσή μου ασχολείται με τη βελτίωση της ασφαλείας των κρατών και των πολιτών στα πλαίσια της δημοκρατικής διακυβέρνησης, ε, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε βάση στη Γενέβη, αλλά έχουμε ένα γραφείο και εδώ στις Βρυξέλλες. Και στη Σλοβενία, την Τινησία, την Παλαιστίνη, το Λίβανο και θα ανοίξουμε και στη Γουατεμάλα ένα γραφείο τους επόμενους μήνες. Συνεργαζόμεθα με τα κράτη-μέλη, ε, με συνεργαζόμενα κράτη, 50 κράτη και διεθνείς οργανισμούς για να στηρίξουμε τα κράτη αυτά και να βελτιώσουμε την διακυβέρνηση τη ασφάλεια μέσω συμμετοχών που, όπως μέσω μεταρρυθμίσεων όπως συμμετέχουν όλοι. Και δημιουργούμε πρωτότυπα προϊόντα, γνώσεις, ε, προωθούμε προδιαγραφές και τις βέλτιστες πρακτικές και βοηθάμε για να αναπτυχθούν οι δυνατότητες ε, στον τομέα της ασφάλειας και για μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Ποια προγράμματα έχουμε με την Ένωση. Πρόσφατα κερδίσαμε ένα διαγωνισμό για την ε, διακυβέρνηση του τομέα της ασφάλειας και βοηθάμε τις αντιπροσωπείες της Ένωσης για το πώς μπορούν να βοηθήσουν τις επιπτώσεις των διαδικασιών διακυβέρνησης της ασφάλειας σε χώρες με τις οποίες συνεργάζονται παγκοσμίω. Επίσης, τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων και η Ένωση μαζί μας ζήτησαν να παίξουμε πιλωτικό ρόλο για το πρόγραμμα για την ε, ε, ενοποιητική διακυβέρνηση της εσωτερικής ασφάλειας. Είναι μια συνεργασία μεταξύ αστυνομικών αρχών που θα ήταν αδιανόητη στα Δυτικά Βαλκάνια πριν από μερικά μόλις χρόνια. Λοιπόν, τι κάνουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες ε, του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων. Πολύ σημαντικό θέμα για την οργάνωσή μας, γιατί δημοσιεύσαμε ένα εγχειρίδιο για αυτό το θέμα πριν από 10 χρόνια. Διαπίστωσα ότι στις 15 Μαΐου 2008 δημοσιεύτηκε αυτό το εγχειρίδιο. Λοιπόν, καλή επέτειος για να συζητήσουμε για αυτό το εγχειρίδιο. Όταν ε, εκπονούσαμε αυτό το πρόγραμμα, θέλαμε να έχουμε κάτι που να περιγράφει τα ανθρώπινα δικαιώματα του προσωπικού ενόπλων δυνάμεων σε ένα κείμενο. Γιατί δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Οπότε αποφασίσαμε να το συγγράψουμε στα πλαίσια της συνεργασίας με τον ΟΑΣΕ αλλά έχει να κάνει και με την Ένωση γιατί έχετε 28 κράτη-μέλη που είναι μέλη του ΟΑΣΕ άρα τα πορίσματά μας ε, έχουν σημασία και για σας ένα από τα κύρια σημεία που αναφέρουμε στο εγχειρίδιο είναι ότι υπάρχουν ε, ε, κατά ανάγκη περιορισμοί των δικαιωμάτων του στρατιωτικού προσωπικού γιατί έχουν ε, ένα ειδικό καθεστώς, μια ειδική θέση στην κοινωνία μας. Υπάρχουν κάποια περιορισμοί λοιπόν, που είναι σημαντικοί για να διατηρηθεί η ασφάλεια και σταθερότητα, ιδιαίτερα σε περιόδους ε, συγκρούσεων. ή σε κάποιες τέτοιες υβριδικές καταστάσεις όπου δεν είμαστε ακριβώς σε σύραξη αλλά υπάρχει εσωτερική αστάθεια για παράδειγμα συγκρούσεις όπως θα δείτε στην ε, παρουσίασή μου δεν είναι ομοιογενής πλήρως ε, η προσέγγιση μας για το θέμα αυτό. Αυτό έχει και θετικά και αρνητικά. Επιτρέπει σε κάθε κράτος μέλος να σχεδιάσει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τους στρατιωτικούς. Όπως είπε και Μάνιολ, πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή μεταξύ των κοινωνικών αξιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ε, αναφερέτων δικαιωμάτων όλων των πολιτών κάποιοι εκ των οποίων είναι στρατιωτικοί. Χρειάζεται λοιπόν να επιτύχουμε αυτή τη χρυσή τομή σε κάθε κράτος. Αυτό όμως ε, δημιουργεί ανισορροπία όταν υπάρχουν ε, διεθνείς επιχειρήσεις, όπως της Ένωσης, όπως των Ηνωμένων Εθνών, του ΝΑΤΟ. Γιατί οι διάφορες στρατιωτικοί έχουν διαφορετικά δικαιώματα, ενώ δουλεύουν ο ένας πλάι στον άλλον. Επιχειρούν ο ένας πλάι στον άλλον, στρατιωτικά. Θα επανέλθω. Τώρα να πω κάτι που είναι αυτονόητο, αλλά θα το πω. Τα ανθρώπινα δικαιώματα των στρατιωτών είναι σημαντικά, όπως τα δικαιώματα όλων των πολιτών. Και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των στρατιωτικών σημαίνει ότι εντάσσονται στην κοινωνία στρατιωτική και ότι δεν είναι ένα χωριστό κομμάτι. μέσω της παροχής αυτών των δικαιωμάτων στους στρατιωτικούς θεωρούμε ότι θα σέβονται αυτά τα δικαιώματα όταν είναι σε επαφή με πολίτες μη στρατιωτικούς σε κάθε κράτος. Αν αρνηθούμε στους στρατιωτικούς τα ανθρώπινα δικαιώματα, άρα δεν θα σέβονται τα δικαιώματα και των υπολείπων πολιτών όταν είναι σε επαφή μαζί τους. Άρα είναι σημαντικό να έχουν ε, παρόμοια δικαιώματα με τους ε, πολίτες. Βέβαια με κάποιους περιορισμούς οι στρατιωτικοί. Το είπα ήδη. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα των στρατιωτικών. Δύο πρότυπα δηλαδή. Το θεσμικό μοντέλο και το εργασιακό μοντέλο. Η διαφορά είναι σε τι βαθμό περιορίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάποιε ε, χώρε θεωρούν ότι πρέπει να είναι πολύ διαφορετικά τα δικαιώματα των στρατιωτικών από των υπολείπων. Αυτό είναι το θεσμικό μοντέλο. Βασίζονται στην προσέγγιση ότι οι ένοπλε δυνάμει είναι μοναδικού χαρακτήρα θεσμό. Εντελώ διαφορετικό θεσμό από του υπόλοιπου θεσμού. Άρα δεν ισχύουν οι ίδιε προδιαγραφέ. Και στηρίζουν, ώστε προωθούν αυτό το μοντέλο, ότι πρέπει να είναι αποτελεσματική ε, και σε ετοιμότητα στρατιωτική ανά πάσα στιγμή. Κάτι που ισχύει και να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται πειθαρχία, στρατιωτική πειθαρχία. Είναι το πρώτιστο. Και αυτό διασφαλίζεται μέσω της ιεραρχικής διοίκηση, για να λαμβάνονται ταχαίω οι αποφάσεις με βάση της ε, κρίσεις του διοικητή. Άλλα κράτη θεωρούν ότι δεν είναι τόσο μεγάλε διαφορέ. Αυτό είναι το επιχειρησιακό μοντέλο, το επαγγελματικό μοντέλο. Θεωρεί το επαγγελματικό αυτό μοντέλο ότι ε, είναι ένα επάγγελμα όπω τα άλλα και πρέπει να ισχύουν τα συνήθη κίνητρα, για παράδειγμα μονιμότητα, μισθή κτλ. Και εδώ θεωρούν ότι πρέπει να δίδονται περισσότερα δικαιώματα. Ιδιαίτερα επειδή οι στρατιωτικοί όλο και πιο πολύ προσεγγίζουν αυτό το επαγγελματικό μοντέλο διότι όλο και πιο πολύ απομακρυνόμεθα από τους κληρωτούς και περνάμε σε επαγγελματικό στρατό. Υπάρχουν περιορισμοί, βεβαίως, αλλά αυτοί οι περιορισμοί δεν μπορεί να είναι αυθαίρετοι. Πρέπει να πληρούν αυτά τα πέντε κριτήρια που βλέπετε εδώ. Πρώτον, πρέπει να βασίζονται σε στρατιωτικές ανάγκες. Δεύτερον, πρέπει να βασίζονται σε νόμους. Πρέπει να είναι ανάλογες με τις ανάγκες. Τέταρτον, δεν θα πρέπει να δημιουργούν διακρίσεις και οποιοδήποτε περιορισμοί που δημιουργούν διακρίσεις πρέπει να αιτιολογούνται σαφώς. Και τέλος, οι ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει να είναι αυτοί που καθορίζουν την ανάγκη αυτούς τους περιορισμούς και όχι κάποιος άλλος. Να αποδεικνύουν αυτούς τους περιορισμούς. Πρέπει όλα αυτά να βασίζονται σε διεθνές δίκαιο. Αν και σε ένα βαθμό προέρχονται και από το εθνικό δίκαιο. Είναι ουσιώδης πηγή. Αλλά κυρίως θα ασχοληθούμε με τις ε, επόμενες αρχές, την διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη Διεθνή Σύμβαση για τα πολιτικά και θεμελιώδη δικαιώματα και το Σύμφωνο των ΗΠΑ για τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, την Σύμβαση των Εθνών κατά των βασανιστήριων, την ε, ε, Σύμβαση κατά των διακρίσεων κατά των γυναικών και άλλες διεθνείς συμβάσεις. Αυτή θα είναι η βάση μας. Οπότε, συγκεκριμένα δικαιώματα τώρα. Δεν θέλω να εστιάσω υπερβολικά σε πολιτικά δικαιώματα. Γιατί αυτά σε μεγάλο βαθμό είναι δικαιώματα που ασκούνται εντός του κράτους μέλους και όχι κατά τη διάρκεια αποστολών στο εξωτερικό. Αλλά παρόλα αυτά έχουν τη σημασία τους. Αυτά τα δικαιώματα πρέπει φυσικά και αυτά να ισχύουν. Λοιπόν, ποια είναι τα δικαιώματα τα βασικά αυτά. Το δικαίωμα να συμμετέχει κανείς σε ένα πολιτικό κόμμα, να εκλέγεται, δικαίωμα έκφρασης, δικαίωμα συνεταιρίζεστε, αντιρρησίες συνείδησης και ελευθερία θρησκευτικής πίστης σε πολλές χώρες. Ο στρατός πρέπει να είναι πολιτικά ουδέτερος και να μην συμμετέχει σε επίμαχα πολιτικά θέματα. Αλλά άλλες χώρες έχουν άλλη προσέγγιση. Θεωρούν ότι οι στρατιωτικοί είναι απλώς πολίτες, ένστολοι πολίτες, όπως είπε και ο Εμάνιελ. Αυτή η διαφορά, αυτή η διάκριση μάλλον, όσοι θεωρούν ότι οι στρατιωτικοί είναι ένστολοι πολίτες, που είναι οι περισσότερες, οι χώρες αυτές δεν περιορίζουν ιδιαίτερα τα πολιτικά δικαιώματα του, των στρατιωτικών. Παρ' όλα αυτά, όλες οι χώρες συμφωνούν ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί των πολιτικών δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών των στρατιωτικών. Αλλά όλα αυτά βεβαίω ε, δεν θα πρέπει να παραβιάζουν τι αρχέ τη ισότητα των μη διακρίσεων και των ίσων ευκαιριών. Υπάρχουν κάποιε κατηγορίε διακρίσεων ε, εθνοτικέ, ε, φύλου, γλωσσικέ και προσωπικό ΛΟΑΔ. Όλες οι συμβάσεις απαγορεύουν τις διακρίσεις με βάση φύλο, χρώμα, θρησκεία, θρησκευτική πίστη κτλ. Αυτή είναι η σύμβαση για τα πολιτικά δικαιώματα που απαγορεύει τη διάκριση κατά εθνοτικών, γλωσσικών και θρησκευτικών μειονοτήτων. Επίσης, προτείνουν ότι πρέπει να γίνει προσπάθεια για να σταματήσουν διακρίσεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, έχει λάβει ενεργά μέτρα για να στηρίξει την κατάργηση των διακρίσεων. Βεβαίω και δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσει και σε βάρο των γυναικών. Γιατί οι γυναίκε είναι πάνω από το μισό του πληθυσμού και υπο-εκπροσωπούνται μονίμως στι ένοπλε δυνάμεις. Πρόσφατα, πολλοί, πολλοί από τους φραγμούς, τους ε, θεσμικούς φραγμούς στη θεωρία για, κατά των γυναικών έχουν ε, καταργηθεί, αλλά εξακολουθεί στην πράξη να υπάρχει διάκριση. Τα κράτη-μέλη πρέπει να εξετάζουν συνεχώ και την ομοθεσία και τι πολιτικέ και τι πρακτικέ του για να μην υπάρχει στην πράξη διάκριση κατά των γυναικών χωρί στρατιωτική αναγκαιότητα. Πολλά κράτη έχουν αρχίσει να αναθεωρούν ενεργά την πολιτική του και με πιο ενεργό τρόπο στρατολογούν γυναίκε. Το ίδιο και για ε, τα άτομα ΛΟΑΔ. Αυτό είναι ακόμη επίμαχο θέμα για πολλά κράτη, σε πολλά κράτη, για πολλά έτη, σε πολλά κράτη, άτομα ΛΟΑΔ εξαιρούντο από τις ένοπλες δυνάμεις σε πολλά κράτη. Μέλη δεν υπάρχει πλέον επίσημη απαγόρευση, αλλά υπάρχουν πολλοί διαρθρωτικοί φραγμοί, όπως και για τις γυναίκες, για το προσωπικό ΛΟΑΔ, ούτως ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει πλήρω στις ένοπλες δυνάμεις. Πρέπει να ληφθούν μέτρα για να μην υπάρχουν άτυποι φράγμη όταν καταργούνται οι τυπικοί φραγμοί. Τώρα θέματα της ζωής στους στρατώνες και γενικότερα της στρατιωτικής ζωής για να μην υπάρχουν ε, ε, να μην υπάρχει κάκο μεταχείριση του προσωπικού. Για παράδειγμα δεν πρέπει να υπάρχουν καψόνια και άλλες μορφές ε, τελετών μοίησης και δεν πρέπει να φτάνει στο άκρο η ανάγκη τήρηση τη πειθαρχία. Για παράδειγμα, δεν πρέπει να επιβάλλεται πειθαρχία με βία μέσα. Και δεν θα πρέπει σε καιρό ειρήνη να γίνεται εξομοίωση μαχών. Δεν πρέπει, για παράδειγμα, να γίνεται ε, υποσυτισμός του προσωπικού για να εξομοιούνται οι συνθήκες πολέμου. Και πρέπει να υπάρχουν οι αναγκαίες εγγύησεις. Η κακομεταχείριση πρέπει να αντιμετωπίζεται να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής των στρατιωτικών που θεωρούν ότι έχουν γίνει αντικείμενο κακομεταχείρισης. Θα πρέπει να υπάρχει διαδικασία δηλαδή υποβολής παραπώνων για όλους τους στρατιωτικούς. Όταν ε, παραβιάζονται τα δικαιώματά τους δηλαδή να έχουν το δικαίωμα να απευθυνθούν σε κάποιο φορέα. Και οι συνθήκε εργασία επίση είναι αρκετά σημαντικό θέμα για το θέμα αυτό. Πρέπει να υπάρχουν ε, επαρκείς ε, συνθήκες διαβίωσης για την ε, προστασία της φυσικής και πνευματικής τους υγείας. Πρέπει να ισχύουν και στους στρατώνες και όταν συμμετέχουν σε αποστολές στο εξωτερικό. Ισχύει ιδιαίτερα για το προσωπικό των όπλων δυνάμεων <clears throat> για να έχουν υψηλό επίπεδο περιβάλλον, ε, υψηλού επίπεδου περιβάλλον εργασίας να αποφεύγονται τα ατυχήματα. Αυτό βελτιώνει και την αποτελεσματικότητα των όπλων δυνάμεων και το πνεύμα ε, ομάδας και βελτιώνει και τη θέση των ενόπλων δυνάμεων στην κοινωνία. Υπάρχουν ανισορροπίες μεταξύ των ε, χωρών που συμμετέχουν σε πολυεθνικές ε, αποστολές και αυτό μπορεί να έχει αντίστροφα αποτελέσματα. Αν υπάρξουν πολλά ατυχήματα, πολλές ασθένειες, μειώνεται η συνοχή των ενόπλων δυνάμεων και αυτό μειώνει την αποτελεσματικότητά τους. Αν σε ε, μια στρατιωτική μονάδα ένα τμήμα έχει θαυμάσια τροφή, θαυμάσια περίθαλψη κτλ. Γενικά θαυμάσιο περιβάλλον εργασίας που εργάζεται δίπλα σε, ένα άλλο, σε μια άλλη μονάδα από μια άλλη χώρα όπου είναι ανεπαρκής η τροφή και η περίθαλψη και όλα αυτά που δεν λαμβάνει επαρκή επιζώματα, δεν πληρώνεται αρκετά και αναγκάζεται να αντισταθμίσει με διάφορε άλλε δραστηριότητε αυτέ τι ελλείψει, αυτό μειώνει την αποτελεσματικότητα τη ίδια τη επιχείρηση. Και αναπόφευκτα οι στρατιωτικοί αυτών των διεθνών αποστολών συγκρίνουν τις συνθήκες τους, ε, την τροφή τους, τα άλλα δικαιώματα των οποίων απολαμβάνουν με, άλλα, με άλλους στρατιωτικούς από άλλες χώρες που συμμετέχουν στην ίδια επιχείρηση. Και αυτή η σύγκριση διαβρώνει την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας. Άρα πρέπει να εξετάσουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την ανισορροπία μεταξύ των εθνικών συνιστοσών μιας πολυεθνικούς συνισταμένης. Πολυεθνικής. Αυτά είναι τα δικαιώματα λοιπόν και αυτές είναι οι επιπτώσεις της στήριξής τους. Και τώρα θέλω να μιλήσω για τους ε, μηχανισμούς ε, επιβολής αυτών των δικαιωμάτων. Πρέπει να υπάρχουν κοινέ προδιαγραφές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά πρέπει να υπάρχουν και κοινέ προδιαγραφές για την ε, άσκηση και προστασία αυτών των δικαιωμάτων. Πρέπει λοιπόν να κωδικοποιηθούν τα δικαιώματα και οι πολιτικές, αλλά πρέπει να παράσχουμε και τους αναγκαίους μηχανισμούς επιτήρησης που θα διαπιστώνουν ότι τηρούνται αυτά τα δικαιώματα και αν δεν τηρούνται πρέπει να υπάρχουν αναγκαίοι μηχανισμοί για να αντιμετωπιστούν αυτές οι παραβιάσεις. Το πρώτο που είναι προληπτικό, να υπάρχει σωστή κατάρτιση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλα αυτά τα δικαιώματα δεν έχουν καμία σημασία εάν το στρατιωτικό προσωπικό δεν τα γνωρίζει. Δεν γνωρίζει τι πρέπει να σέβεται. Πρέπει να υπάρχει τακτική κατάρτιση όλου του στρατιωτικού προσωπικού για τα θέματα αυτά. Για να προλάβουμε και παραβιάσεις τους όταν ε, συμμετέχουν σε αποστολές στο εξωτερικό. Πέρα από το, την νομοθεσία πρέπει να υπάρχουν και κώδικες δεοντολογίας, επαγγελματικοί κώδικες ε, σωστής ε, συμπεριφοράς. Και βεβαίως και στις ε, στρατιωτικές σχολές πρέπει να διδάσκονται αυτά τα δικαιώματα. Έτσι διασφαλίζουμε ότι ο σεβασμός είναι βασικό στοιχείο της εκπαίδευσης όλων των αξιωματικών σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας. Εφόσον λοιπόν γνωρίζουν στρατιωτικοί τα δικαιώματα, αυτά πρέπει κατόπιν επίσης να ελέγχονται και για ενδεχόμενε παραβιάσει αυτών των δικαιωμάτων. Η στρατιωτική αποτελεσματικότητα βασίζεται στην ε, τήρηση κανόνων και διαταγών. Και εφόσον ε, η τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι τμήμα αυτών των κανόνων, πρέπει και αυτοί να γίνονται σεβαστοί. Οι διοικητέ λοιπόν είναι υπεύθυνοι όχι μόνο για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και για να δρούν ταχαίω και αποτελεσματικά για να ε, διασφαλίζουν αυτή την τήρηση. Πρέπει να έχουν υπόψη οι διοικητές ότι είναι οι πρώτοι αρμόδιοι για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην μονάδα τους. Πρέπει λοιπόν να έχουν την αναγκαία πείρα, αλλά να γίνονται και σεβαστοί για να τηρούνται και οι διαταγές που δίνουν γι' αυτό. Βεβαίως, ο στρατός πρέπει να εκτελεί διαταγές. Αλλά κάθε στρατιωτικό είναι υπεύθυνο για τη συμπεριφορά του. Εάν κάνει κάτι παράνομο, είτε αυτοβούλο είτε κατόπιν διαταγή, πρέπει κατόπιν να ελεγχθεί. Είναι σημαντικό να υπάρχουν οι αναγκαίε διατάξει για να προστατεύονται οι στρατιώτες που αρνούνται να εκτελέσουν παράνομες διαταγές εάν τους δοθούν. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, η ιεραρχική δομή μπορεί να επιλύσει ταχαίως τα περισσότερα προβλήματα. Η ιεραρχία δηλαδή. Αν δεν συμβεί όμως αυτό, σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να στραφούμε προς τα πολιτικά δικαστήρια ή τα στρατοδικεία. Εάν λειτουργεί το σύστημα της στρατιωτικής δικαιοσύνης που έχει το στόχο να διασφαλίσει την εφαρμογή της πειθαρχία και επίσης την εφαρμογή του δικαίου. Όλα τα ε, πειθαρχικά θέματα μπορούν να επιληθούν από τους διοικητές. Αλλά ορισμένα δεν μπορούν να επιληθούν, τότε πρέπει να απευθυνθούμε στι αρμόδιες αρχές που μπορεί να είναι στρατιωτικού ή πολιτικού χαρακτήρα. Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις για, για τα συστήματα στρατιωτικής δικαιοσύνης εάν πρέπει να υπάρχουν ειδικευμένα στρατιωτικά δικαστήρια ή εάν τα πολιτικά δικαστήρια μπορούν να αποδώσουν δικαιοσύνη για τους στρατιωτικούς. Αυτό είναι ακόμη θέμα συζήτησης. Αλλά απομακρυνόμεθα όλο και περισσότερο από τα στρατοδικεία και προσεγγίζουμε όλο και περισσότερο την υπαγωγή των ε, υποθέσεων αυτών στα πολιτικά δικαστήρια. Θα πρέπει να τελειώνεται ο Σονούπο. Θα πρέπει να τελειώνεται ο Σονούπο. Βεβαίω. Σε ό,τι αφορά την στρατιωτική δικαιοσύνη, υπάρχουν δύο τομεί ανησυχία. Καταρχά, ε, το θέμα τη ανεξαρτησία του συστήματο στρατιωτική δικαιοσύνη και το, το δικαίωμα σε μια δίκαιη δική. Για να θεωρείται αξιόπιστη η στρατιωτική δικαιοσύνη, θα πρέπει να απομακρυνθεί από την στρατηγική διοίκηση, γιατί υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα σε αυτού που, κάνουν, που υποβάλλουν μια αγωγή και σε αυτούς που κρίνουν την αγωγή. Σε ό,τι αφορά το θέμα της δίκης δίκης τα μέλη του στρατηγικών δυνάμεων θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως και οι πολίτε στο βαθμό του δυνατού. Αυτό αφορά την πρόσβαση σε νομικέ συμβουλέ και εκπροσώπηση ε, στην επιβολή μας της πειθαρχίας το στρατιωτικό σύστημα δικαιοσύνης θα πρέπει να σέβεται και τα δικαιώματα σε μια δική δίκη ε, και το δικαίωμα αυτό ε, συνδέεται άρρηκτα με την ανεξαρτησία των στρατιωτικών δικαστηρίων. Το τελευταίο, τελευταίο σημείο που έχω για το μηχανισμό υποπτίας είναι για δημοσιολάβηση και φορείς δημοσιολάβησης θεσμούς εθνικούς για τα δικαιώματα, κοινοβουλευτικούς επιτρόπους κλπ. Αυτοί οι θεσμοί που σημαντική φορεί στην παροχή της στρατιωτική δικαιοσύνης και ότι το σύστημα λειτουργεί εύρυθμα και είναι αποτελεσματικότερο και δεν δημιουργεί προβλήματα. Και θα πρέπει αυτοί οι δημοσιολαβητές να εποπτεύουν το σωτικό τομέα, εξετάζοντα καταγγελίε και προστατεύοντα τα ανθρώπινα δικαιώματα και αποφεύγοντα την μη χρηστή διαχείριση. Αυτή η διαμεσολαβητική φορεί θα πρέπει να είναι εξάρτητη από τη διοίκηση. Έτσι μπορούν να ασκήσουν την εποπτεία τη στρατιωτική δικαιοσύνη και του συστήματο και του στρατιωτικού τομέα χωρί να επηρεάζονται από τη δίκηση. Αυτή η εποπτεία είναι πολύ απαραίτητη. Μπορούν να εντοπιστούν συστημικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο στρατιωτικό τομέα και να δίνονται συστάσει για την μεταρρύθμιση των προβληματικών τομέων. Χωρίς αυτή την ανεξαρτησία και την ε, εικόνα ανεξαρτησίας δεν θα είναι αποτελεσματικοί οι φορείς διότι δεν θα εξυπηρετούν ε, ένα σκοπό που είναι διαφορετικός από το, από το δικαστικό, το μεσοτικό Και επίσης οι δημοσιολαβητικοί φορείς ε, μπορούν να επιλύουν τα προβλήματα, να διενεργούν έρευνες που είναι εναλλακτικό τρόπο προστασία των ατόμων από άδικε αποφάσει, παραβιάσει των δικαιωμάτων αυτών ή κατάχρηση εξουσία. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι δημοσιολογητικοί φορεί δεν αντικαθιστούν τη στατιωτική δικαιοσύνη, τα στατοδικεία και οι δημοσιολογητικοί φορεί δεν αντιμετωπίζουν ποινικέ υποθέσει, αλλά εξετάζουν καταγγελίε όσον αφορά παραβιάσει δικαιωμάτων λόγω διαχείριση διαχείρισης. Τα σοβαρά ποινικά δικήματα πάντα αντιμετωπίζονται από τα πολιτικά, τα δικαστήρια, τα στατοδικεία. Και οι δημοσιολαβητικοί φορεί έχουν δυνατότητα επιβολή των μέτρων και εξαρτώνται από την πιστοσύνη ε, των συστάσεων που κάνουν οι στερετικοί ή τα κοινοβούλια που ελέγχουν τη δραστηριότητά τους. Τούτων λεκθέντων υπάρχουν κάποιες τάσεις εντός των δικαιωμάτων του στερετικού προσωπικού τα τελευταία χρόνια. Πρώτη τάση είναι ότι ο στρατιωτικό τομέα, το στρατιωτικό προσωπικό αποτελεί περισσότερο από επαγγελματίε, δεν έχουμε πλέον κληρωτούς τόσου πολλού. Σαν αποτέλεσμα αυτού, οι στρατιωτικοί πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια τόσο ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι συνθήκες ε, της υπηρεσίας ε, είναι πιο ελκυστικές για να μπορούν να ανταγωνιστούν άλλους εργοδότες στην αγορά. Αυτό συνεπάγεται αύξηση των ευεργετημάτων όπως είναι οι πληρωμές, η υγειονομική περίθαλψη κυρίως ε, μετά την αποστράτευση και αυτό έχει αντίκτυπο τις ελάχιστες προδιαγραφές των υπηρεσιών που παρέχουν οι ένοπλες δυνάμεις στο προσωπικό τους. Πολύ συχνά οι ένοπλες δυνάμεις ε, εξυπηρετούν μη παραδοσιακούς ρόλους, όχι μόνο σε πολέμους, αλλά σε νευτικές διαδικασίες, ε, που πρέπει να επιβάλλουν την ειρήνη. Δεν πολεμούν μόνο σε πολέμους, αλλά προστατεύουν και την ειρήνη και σε εσωτερική αστυνόμευση, προστασία των συνόρων, ε, παροχή βοηθεία σε περιπτώσεις καταστροφών, και όλα αυτά δημιουργούν διάφορες υποχρεώσεις για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων δεν δεσμεύονται μόνο από το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και τον νόμο για τις ενόπλες συγκρούσεις, αλλά επίσης δεσμεύονται και από διεθνή νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως ανέφερα ήδη, σαν αποτέλεσμα όλων αυτών, πολλοί από τους νέους ρόλους γίνονται όλο και περισσότερο πολυμερείς στη φύση τους, άρα γίνεται και περισσότερη σύγκριση και ρίχνεται φως στις διαφορές που υπάρχουν ε, στις, ε, στα δικαιώματα που έχουν τα διάφορα εθνικά στρατεύματα και αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ηθικό σε, των στρατευμάτων σε διεθνείς αποστολές. Αυτές οι πολυεθνείς αποστολές, οι διεθνείς αποστολές ε, ε, χρειάζονται μεγαλύτερο συντονισμό, χρειάζονται κοινά πρότυπα για να εξασφαλίζεται τη λειτουργικότητα μεταξύ δυνάμεων διαφορών εθνικοτήτων. Αυτό συχνά εστιάζεται επί τεχνικών ζητημάτων, όπως ε, είναι ε, η διάμετρος των σφαιρών ε, και διάφορα τεχνικά ζητήματα και, διάφορα θέματα που αφορούν και τα ανθρώπινα δικαιώματα των ενόπλων δυνάμεων, κάτι που αναφέρθηκε, πρέπει να υπάρχουν κοινά πρότυπα τελικά για τα δικαιώματα του προσωπικού και το πώς ε, να ζητήσουν να δικαιωθούν αν έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά τους. Κάτι τελικό. Μιλάμε για περισσότερα ανθρώπινα δικαιώματα για το προσωπικό των όπλων δυνάμεων και καταπολέμηση των διακρίσεων και ίση εκπροσώπηση των ενόπλων δυνάμεων. Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα οι επικριτές θα έλεγαν ότι κάτι τέτοιο θα υπονόμευε την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των όπλων δυνάμεων δίδοντας τη δυνατότητα στις γυναίκες να υπηρετούν στις αναπλές δυνάμεις. Αυτή ήταν μια σταθερή μακροχρόνια επίκριση, θα υπονομευόταν η αποτελεσματικότητα των ενόπλων δυνάμεων, όταν όμως μετά από την ένταξη των γυναικών στις ενόπλες δυνάμεις η αποτελεσματικότητα δεν υπονομεύτηκε και πολλές μελέτες κατέδειξαν το αντίθετο μάλιστα και αυτή η αποτελεσματικότητα αυξήθηκε. Έτσι, πολλοί από τους επικριτές που δεν θέλουν περισσότερα δικαιώματα στο προσωπικό και ίση εκπροσώπηση στο στρατό, ε, πιστεύω ότι υπερβάλλουν στα επιχειρήματά τους. Η ειδική μέρημνα πρέπει να λαμβάνεται ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη επικρίσεις. Δεν θα γίνει ο στρατός λιγότερο αποτελεσματικός σε θετική, έχουν περισσότερα δικαιώματα. Πρέπει να εξεταστεί περισσότερο. Και πρέπει να καταπολεμηθούν αυτές οι επικρίσεις. Νομίζω ότι έτσι συνοψίζεται η παρουσίασή μου, ολοκληρώνεται η παρουσίασή μου. Και σας ευχαριστώ για την προσοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τους δυο σας ενδιαφέρουσες και λεπτομερείς οι παρουσιάσεις σας. Τώρα ε, θα υπάρξει ανταπόκριση στις εκκλήσεις σας για ερωτήσεις και θα δώσω έτσι το λόγο στους συναδέλφους. Ο Μάικλ Γκάλλερ είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, βεβαίως, ευχαριστώ για την, ε, το γενικό χαιρετισμό που κάνατε στους υπό υπαξιωματικούς της αεροπορίας της Γερμανίας στο Άπελ, στο Σλέσφι Χολστάιν. Όταν έρχονται σε εμά, μάλλον όταν έρχονται στις Βρυξέλλες οι στρατιωτικοί, εγώ του λέω πάντα να μην πάνε μόνο στο ΝΑΤΟ, αλλά να έρθουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι σημαντικό θεσμό. Θα πρέπει να έχουμε περισσότερε τέτοιε επισκέψει από στρατιωτικού στην Επιτροπή μα. Πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Γιάγκομπ, επειδή ήμουνα εισηγητή για την Ουκρανία. Πρέπει να πάω κάπου αλλού, δεν άκουσα την αρχή τη ομιλία του, αλλά γνωρίζω τι θέσει του. Και θεωρώ ότι είναι καλή ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Είδαμε πρώτα απ' όλα λοιπόν τα γενικά δικαιώματα των στρατιωτών ως πολιτών. Είναι φυσιολογικό βεβαίως ε, να εφαρμόζονται με συγκεκριμένο τρόπο στην υπηρεσία και ιδιαίτερα όταν έχουμε αποστολές πολυεθνικός της Ένωσης. Είναι σημαντικό να μπορούν να εκφραστούν ακριβώς οι στρατιωτικοί, να μας πούν τι ανεπάρκειες υπάρχουν, τόσο ώστε εμείς να ενημερωθούμε ως πολιτικοί και να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Στο παρελθόν, και σε κάποιες χώρες ε, εξακολουθεί να υπάρχει κατάσταση όπου δεν επιτρεπόταν ε, η δημιουργία επαγγελματικών ενώσεων και σε κάποιες χώρες είναι μεγάλες οι δυσχέρειες ακόμη. Νομίζω ότι το αναφέρατε αυτό, έτσι δεν είναι. Πρέπει να συζητήσουμε με τους συναδέλφους από τις χώρες αυτές. Θεωρώ ότι στις χώρες που μπορούν να οργανωθούν οι στρατιωτικοί για να προωθήσουν τα συμφέροντά τους αυτό μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία των όπλων δυνάμεων. Και δεν ενοχλεί. Εδώ δεν πρόκειται βέβαια να χορηγήσουμε δικαίωμα απεργία στους στρατιωτικούς όταν πρόκειται να πολεμήσουν. Αλλά πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, ε, για παράδειγμα, αυξήσεις. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Να μην υπάρξουν παρανοήσεις. Οι ερωτήσεις μου λοιπόν είναι οι εξής. Υπάρχει συνειδητοποίηση ότι πρέπει να υπάρξουν κοινέ ρυθμίσει όταν γίνονται κοινέ αποστολέ. Και αν οδεύουμε προ αυτή την κατεύθυνση. Είπατε για παράδειγμα για την περίθαλψη. Υπάρχει ένα πρόγραμμα στα πλαίσια της ΠΕΣΚΟ που επιδιώκει να υπάρξει εναρμόνιση. Να υπάρξει ένα κοινό ιατρικό κέντρο για τις επιχειρήσεις. Οπότε τότε θεωρούμε ότι όταν συμμετέχουν κάποιοι σε μια επιχείρηση, τότε μέσω αυτού του κοινού κέντρου θα έχουν την ίδια περίθαλψη. Αλλά δεν περιορίζεται βέβαια εκεί μόνο το θέμα. Το θέμα είναι τι φροντίδα θα έχουν και κατόπιν. <clears throat> Εφόσον κάποιοι βεβαίως συμμετέχουν σε μια επιχείρηση, μπορεί να υπάγονται στους ίδιους κανόνες. Αλλά κατόπιν, εκ των υστέρων, μπορεί να μην ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι σημαντικό αυτό. Πρέπει να υπάρξει πολιτική λύση. Να μην ε, μειονεκτούν κάποιοι που συμμετέχουν σε μία αποστολή της Ένωσης και αντίστοιχα βεβαίως ε, να μην ε, αντιμετωπίζουν, δηλαδή να αντιμετωπίζουν χειρότερες καταστάσεις κάποιοι σε μία πολυεθνική κατάσταση ε, να αντιμετωπίζουν καταστάσει που θα ήταν χειρότερες από εάν είχαν συμμετάσχει σε μια εθνική αποστολή. Ευχαριστώ Μάικλ. Ο κ. Σεύκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω εγκαρδίω για τις πληροφορίε που μας δώσατε, για τις παρουσιάσεις. Αφετηρία τη συζητήσεω θα έπρεπε να ήταν κατά την άποψή μου η αρχή σύμφωνα την οποία ένας στρατιώτη είναι και ένας πολίτης. Το πρόβλημα οφείλεται στο ότι αν αναλύσουμε την κατάσταση που επικρατεί στα κράτη-μέλη, οι στρατιώτε έχουν πολύ διαφορετικά δικαιώματα. Εγώ εκπροσωπώ την Πολωνία. Στην Πολωνία, όσο ένας στρατιώτης υπηρετεί, δεν μπορεί να συνδικαλίζεται, ενώ ένας αστυνομικός έχει αυτό το δικαίωμα μπορεί να γίνει μέλος ενός συνδικάτου. Ο στρατιώτης δεν μπορεί να είναι μέλος συνδικάτου, δεν μπορεί να είναι μέλος ενός κόμματος και έναντι αυτής της καταστάσεως ο ρόλος των θεσμών ε, ζητεί την ψήφο του στρατιώτου. Ε, ο ρόλος είναι σημαντικό του διαμεσολαβητή στην Πολωνία σε αφορά τα θέματα. Κάτι που δεν εμφανίστηκε στι ε, παρουσιάσει σα και που θεωρώ σημαντικό είναι το εξή. Θα έλεγα και επώδυνο στοιχείο. Οι διαφορέ που υπάρχουν. Υπάρχουν πολύ μεγάλε διαφορέ από χώρα σε χώρα και εντό μια χώρα και είναι επώδυνε οι διαφορέ. Παραδείγματο χάρη, το δικαίωμα που έχει ένα στρατιώτη στη σύνταξη από τη στιγμή που θα προστατευτεί. Το στρατιωτικό του δικαίωμα εξαρτάται από τη στιγμή που ξεκίνησε τη στρατιωτική του σταδιοδρομία. Το 89 έγινε μια επανάσταση στην Πολωνία που ευτυχώς ήταν μια ειρηνική επανάσταση. Εάν κάποιος ξεκίνησε τη στρατιωτική του υπηρεσία πριν το 89 είχε δικαιώματα που δεν έχει αυτός που ξεκίνησε τη θητεία του μετά το 89. Αν πεθάνει κάποιος, ένα, ένα στατιώτης πεθάνει, που συμβαίνει δυστυχώς, δεν έχει δικαίωμα κάποιων παροχών, η οικογένειά του, αν κάποιος τραυματιστεί, έχει κάποια δικαιώματα. Αλλά και εκεί υπάρχει υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Πιστεύω ότι είναι ένα πρόβλημα δεν θα πρέπει να διχάζουμε τους, ε, να διαιρούμε μάλλον τους στατιώτες ανάλογα με την έναρξη της στατιωτικής τους ε, θητείας. Δεν φταίνε αυτή Η ημερομηνία έναρξης στατιωτικής θητείας καθορίζει δυστυχώς τα δικαιώματα που έχουν. Ξέρω ότι η Euromil γνωρίζει το πρόβλημα, το πολωνικό, και θα ήθελα να σας ζητήσω να προσέξετε αυτό το πρόβλημα, διότι αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση κατά την οποία υπάρχουν κατηγορίες στατικών και αξιωματικών συναρτήσει μόνο της ημερομηνία έναρξης της υπηρεσίας τους, Ανάλυση των καθηκόντων τους. Ευχαριστώ κύριε Ζεύκα. Ο κύριος Τρογεύσκη έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ξεκινώντας θα ήθελα να πω ότι εξεπλάγει κάπως διότι ένας από τους συγκεκριμένους είπε ότι δεν θα έπρεπε να το πει, αλλά παρόλα αυτά θα το έλεγε. Και τι είπε. Είπε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, πρέπει να ισχύουν κυρίως και για τους στρατιώτες. Πρέπει να πω ότι μια τέτοια θέση δεν μου φαίνεται και πολύ παρακινδυνευμένη, είναι κάτι φυσικό. Ε, ένας στρατιώτης έχει ακριβώς τα ίδια δικαιώματα όπως κάθε ανθρώπινο όν. Ε, και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να πιστεύει κανείς ότι με τέτοια διαπίστωση μπορεί να συνδέεται με κάποιο κίνδυνο σε μια ομιλία. Αλλάζω θέμα τώρα. Εκείνο που έλειψε από τις παρουσιάσεις σας ήταν πληροφορίες που θα μπορούσαν να δείχνουν τις μεγαλύτερες και πιο ανησυχητικές διαφορές, τις πιο πόδινες διαφορές που υπάρχουν κάποιες διαφορές θα μπορούσαν να μην υπάρχουν. Παράδειγμα, ένας στρατιώτης, Ιταλός, Βρετανός, Πολωνός, συμμετέχει σε μια αποστολή. Θεωρώ προφανές ότι κάθε στρατιώτης θα πρέπει να δέχεται την ίδια διατροφή. Βέβαια υπάρχει και περίπτωση που ένας Ιταλός προτιμάει να φάει ε, πάστα, ενώ ένας Γερμανός προτιμά να φάει λουκάνικα. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα να υπάρχει ένα μενού που θα είναι το ίδιο για όλους. Αλλά πιστεύω ότι κάποιες στοιχές όμως της ε, κάλυψης πρέπει να είναι εναρμονισμένες. Τα εμβόλια, φερειπίν. Αν οι στατιώτες πάνε σε μια αποστολή στην Αφρική, θα πρέπει οι στατιώτες να προετοιμαστούν. Θα πρέπει να προστατευτούν ιατρικά με τον ίδιο ακριβώς ε, τρόπο. Αυτά είναι τα βασικά πρότυπα. Αυτή είναι η βάση για την ασφάλειά τους. Ε, υπήρχαν κάποιες, ε, ε, είδα ποιες εγκαταστάσεις, κάποια στατόπεδα που έμεναν οι στατιώτες και είδα ότι στους, ε, στους καταβλισμούς αυτούς υπήρχαν διαφορές. Κάποιοι εκεί που κοιμόταν μπορούσαν να βάλουν αφήσει και φωτογραφίες, αλλού σε άλλα στατόπεδα οι στρατιώτες άλλων ε, εθνικοτήτων δεν είχαν δικαίωμα ε, διακόσμησης ε, στο χώρο ύπνου. Δεν μπορούσαν να βάλουν τα φύσεις ούτε διακοσμητικά στοιχεία. Θα πρέπει λοιπόν να εντοπιστούν καλά οι διαφορές οι οποίες είναι άδικες και που είναι επώδυνες και δεν θα έπρεπε να εφίστανται. Αυτά και ευχαριστώ. Thank you. Mr. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω ισπανικά. Ευχαριστώ και τους δύο εισηγητές για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσαν. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση προς την εκπρόσωπο της Euromil. Αν η Euromil ξέρει αυτό που συμβαίνει στην Ισπανία για τον νόμο του 2006 ε, για την υποχρεωτική αποστράτευση στρατιωτικών που είναι πάνω, άνω των 45. Αυτό όχι, σημαίνει όχι μόνο απώλεια χρημάτων ε, για τη χώρα μου, αλλά και προφανή ε, διακριτική μεταχείριση ε, εναντί αυτών των ε, στρατιωτών που, είναι υποχρεωτικ... που αποστατεύονται υποχρεωτικά. Εμείς έχουμε πολύ σοβαρά ε, προβλήματα στον Ισπανικό στρατό ε, γιατί υπάρχει σεξουαλική παρενόχληση. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ειδική μονάδα για την παρενόχληση. Ε, επίσης μας απασχολεί η χρήση της θρησκείας στο στρατό. Ε, τιμωρούνται οι στρατιωτικοί που δεν πάνε στην λειτουργία, ας πούμε. ή επίσης ε, θέματα υποστολής της σημαίας Thank you. για θρησκευτικές γιορτές, ενώ θα πρέπει να ανακατέψουμε το θρησκευτικό με το πολιτικό κομμάτι. Δεν θα μιλήσω ως πρόεδρος, αλλά ως ε, απλό μέλος της υποεπιτροπής. Καταρχάς, ε, καλωσορίζω αυτό που είπατε για τα δεντολογικά θέματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα των στρατιωτών θα πρέπει να είναι ένα καθολικό πρότυπο που να αφορά όλους. Σε ό,τι αφορά την υπο... τις ευθύνε και την λογοδοσία που έχει ο καθένας, προφανώς δεν το αμφισβητώ. Δεύτερον, για αυτό που είπε ο Εμμανουέλ, για τις ειδικέ περιπτώσεις ε, για την Ιρλανδία, για την Ιρλανδική υπόθεση. Τι προηγούμενο υπάρχει και τι περιμένετε να ε, υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστούν αυτές οι αποφάσεις ε, ευρύτερα πέρα της Ιρλανδίας. Και τέλος, αυτό που είπατε για το προσωπικό που έχει αποστατευτεί. Τι περίθαλψη τους δίνουμε, τι σύνταξη έχουν, τι επιδόματα έχουν κτλ. Κάτι άλλο που δεν έχετε θίξει είναι ε, το σύνδρομο ε, το μετατραυματικό. δεν θα πρέπει να υπάρχει η ίδια περίληψη σε στρατιωτικό προσωπικό που πλέον έχει αποστρατευτεί. Οι ίδιες παροχές, η ίδια φροντίδα κτλ. Ο Εμμανουέλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους βουλευτές για τις ενδιαφέρουσες παρουσίες τους, παρουσιάσεις τους, ε, τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Κύριε Γκάλερ. Έχω εξηγήσει το, για το δικαίωμα που συνεταιρίζεστε και τη μεγάλη διαφορά που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα κράτη-μέλη. Τεράστιε διαφορέ από κράτος σε κράτος. Θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι είμαστε ευγνώμονες προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι κατ' επανάληψη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε το δικαίωμα αυτό του συνεταιρίζεσαι. Τελευταία φορά ε, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Μηχανισμού. Ε, οργανισμού, συγγνώμη. Και κάτι που είπα και πριν. Πιστεύουμε ότι αυτό το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε, παρότι δεν είναι το βασικό θέμα της ε, συνεδρίασης, είναι τόσο σημαντικό, γιατί χωρίς αυτό, χωρίς ένα ξεκάθαρο σύστημα όπου δεν είναι γνωστό ποιο είναι ο κοινωνικό εταίρο, ε, χωρί να ξέρουμε ποιε είναι οι αρμοδιότητε του κάθε κοινωνικού εταίρου, για να μπορούν οι πολιτικές και θετικές αρχές να δουλεύουν, να συνεργάζονται με τους κοινωνικούς εταίρους για να υπερασπιστούν τα συμφέροντα του στρατιωτικού προσωπικού, είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε. Επίσης, σε άλλες ερωτήσεις σας είπατε ότι δεν υπάρχει το δικαίωμα ας πούμε, στην Πολωνία να ανήκει κανεί σε ένα συνδικάτο. Δεν υπάρχουν πολιτικά δικαιώματα, αν και δεν το συζητάμε αυτό σήμερα, έτσι, τα πολιτικά δικαιώματα. Όταν εξετάσαμε την Πολωνία, η Πολωνία έχει ένα εσωτερικό δικό της σύστημα, όπου το στρατιωτικό προσωπικό εκπροσωπείται από μια ένωση, η οποία εργάζεται εσωτερικά, εντός δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων. Υπάρχουν πολλές τέτοιες ενώσεις και μπορεί κανείς να επιλέξει να ανήκει σε μια ένωση ανάλογα με το βαθμό του. Έχεις ε, ενώσεις για αξιωματικούς και μη αξιωματικούς. Δεν θέλω τώρα να εστιάσω στην Πολωνία. Όταν εξετάζω όμως, βλέπω την πολωνική κατάσταση, συνειδητοποιώ ότι μόνο η ένωση των αξιωματικών μπορεί να αντιμετωπίσει, μπορεί να μιλήσει με τον Υπουργό ε, ή με τον ε, ΓΕΘΑ, Αρχηγό ΓΕΘΑ. Ε, αν υπάρχει πρόβλημα με τους υπαξιωματικούς, ας πούμε, έβλεπα, ε, θεωρώ ότι ο υπαξιωματικό μπορεί να, να σκοτωθεί για τη χώρα του, αλλά δεν έχει το δικαίωμα να μιλήσει, ας πούμε, με τον Υπουργό Άμυνας. Θεωρούνται πολύ κατώτεροι, ας πούμε, για να μιλήσουν με τον ε, Υπουργό. Δεν λειτουργεί αυτό το σύστημα. Γι' αυτό προωθούμε ανεξάρτητες ενώσεις και συνδικάτα που εκπροσωπούν όλο το στρατιωτικό προσωπικό. Κύριε Γκάλε, Φυσικά δεν μιλάμε για το δικαίωμα στην απεργία. Πάντα επανέρχεται σε αυτή τη συζήτηση για τα δικαιώματα των στρατιωτών, το θέμα του δικαιώματος απεργίας. Δεν μπορούμε να φανταστούμε, ας έναν στρατιωτικό ή ένα στρατιώτη να απεργεί, έτσι. Στην Ευρώπη, ε, σε ορισμένα κράτη, έχουμε συνδικάτα που κάνανε ας πούμε, μισάωρη απεργία. Έχουμε, ας πούμε, εδώ στο Βέλγιο, ε, διαδηλώσεις Βλέπουμε, βλέπουμε ένστολους, πούμε, αλλά χωρίς σημαίες κτλ. Ή στην Ελισσαβόνα α πούμε, το περασμένο Σαββατοκύριακο έγινε μια διαδήλωση και στην Ισπανία, μάλιστα. Ε, με όλα αυτά τα προβλήματα που μα αναφέρατε στην Ισπανία. Αλλά διαδηλώσει γίνονται, αλλά ποτέ απεργία στην Ευρώπη των στρατιωτικών, του στρατιωτικού προσωπικού. Έτσι. Επίσης, για την υπόθεση Γιουρομήλ αντίον Ιρλανδίας, για την χάρτη των κοινωνικών δικαιωμάτων. Η Euromillan είπε ότι, ή μάλλον το δικαστήριο είπε ότι είχε άδικο η Ιρλανδία που δεν δίνει τα δικαιώματα κοινωνικά δικαιώματα στους στρατιωτικούς, αλλά φυσικά με βάση την απόφαση αυτή δεν έχουν το δικαίωμα στην απεργία, έτσι, το στρατιωτικό προσωπικό. Για το ερώτημα του κ. Γκάλε, για την κοινή προσέγγιση σε επιχειρήσεις, ε, την ε, κοινή ιατρική περίθαλψη και αν υπάρχει πρόοδος σε αυτό το μέτωπο. Ναι, υπάρχει όλο και περισσότερο, αλλά δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι προχωράμε λόγω του ότι στον ιατρικό τομέα τα κράτη δεν έχουν τη δυνατότητα από μόνα τους να δώσουν ε, όλη την ιατρική περιθάλψη που χρειάζονται οι στρατιώτες. Έχουμε όλο και περισσότερο διάφορες χώρες που είναι, ή μία χώρα που είναι υπεύθυνη για την ιατρική περίθαλψη. Το θέμα δεν είναι ποια χώρα είναι υπεύθυνη για την ιατρική περίθαλψη κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Τι γίνεται όταν τα άτομα αυτά επιστρέψουν στη χώρα τους, όταν δεν είναι πια στην αποστολή, στην επιχείρηση και όταν επιστρέψουν στη χώρα και αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της επιχείρησης. Γιατί εκεί εντάσσονται εκ νέου στο εθνικό πλαίσιο. Και σε ορισμένα κράτη-μέλη η ιατρική περίθαλψη είναι θαυμάσια. Οι κοινωνικοί φροντίδα σε περίπτωση που έχουμε τραυματία στρατιώτη ή κάποιο στρατιώτη που πεθαίνει. Η περίθαλψη που δίνουν οι, οι ένοπλες δυνάμεις ε, στο προσωπικό τους δεν αφορά μόνο το τι κάνει η καρδιά και της του ο στρατιωτικός ή ο στρατιώτης. Τι το βασικό θέμα είναι τι γίνεται αυτή τη στιγμή ή αποστατευτεί ή αυτή τη στιγμή μείνει μόνη τη η χείρα του. Επομένω, θα πρέπει να συντονιστούμε και να φτάσουμε σε ένα νέο επίπεδο για το τι συμβαίνει μετά την αποστολή, την επιχείρηση. Ευχαριστώ και τον Πολωνό μιλητή που δέχεται ότι και οι στρατιώτες είναι πολίτες, απλώς φοράνε μια στολή. Ε, και τα διάφορα δικαιώματα στα κράτη-μέλη αναγνωρίζει ότι δεν είναι στο ίδιο επίπεδο και υπάρχει πρόβλημα. Επανήλθαμε στο θέμα των συνδικάτων ή των ενώσεων στην Πολωνία, το συζητήσαμε. Το πρόβλημα που αναφέρατε είναι η συζήτηση για το σταξιδοτικό στην Πολωνία. Την ξέρουμε αυτή τη συζήτηση και προσπαθούμε να την παρακολουθήσουμε. Είμαστε σε επαφή με τις οργανώσεις μας στην Πολωνία και με τον διαμεσολαβητή για τα ανθρώπινα δικαιώματα που εξετάζει αυτό το θέμα και παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά και αυτό που κάνετε εδώ στο Κοινοβούλιο και αυτό που κάνετε πρόσφατα για το θέμα αυτό. Να. Επανέλθω λιγάκι στο πώς ε, το προσωπικό μας εκπροσωπείται στις ε, πολωνικές ενόπλες δυνάμεις. Και εκεί βλέπουμε να υπάρχει πρόβλημα. Οι ενώσει που θα πρέπει να υπρασπίζονται το στρατιωτικό προσωπικό το κάνουν τον καλύτερο τρόπο, γιατί εξαρτώνται κατά μεγάλο βαθμό από την καλή θέληση της ε, κυβέρνησης ή των ε, νόπλων δυνάμεων. Επομένως, ε, μπλοκάρει στροποντινά αυτούς που εκπροσωπούν το, τους στρατιώτες. Πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί είναι απαράδεκτο το στρατιωτικό προσωπικό και το δικό σας στρατιωτικό προσωπικό τόσα χρόνια μετά χωρίς κάποιος να έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα, να χάνει ας πούμε ένα τμήμα της σύνταξή του ή όλη τη σύνταξή του γιατί απλώς ας πούμε ξεκίνησε την θητεία του κάποια συγκεκριμένη στιγμή κτλ. Δεν θα σας βοηθήσει τώρα, δεν θα σας καθησυχάσει, δεν θα σας παρηγορήσει το γεγονός ότι δεν είσαστε μόνοι. Εδώ και στην Τσεχία το ίδιο προβλήματα έχουμε. Εδώ και πολλά χρόνια προσπαθούμε να ξανοίξουμε τη συζήτηση, αλλά δεν το θέλουν. δεν το θέλει η σημερινή κυβέρνηση της Τσεχίας αυτό, το να συζητήσει αυτά τα θέματα. Ανθρώπινα δικαιώματα για τους στρατιώτες. Φυσικά, είναι κάτι λογικό και κατά γνώμη μας. Αλλά βλέπουμε ότι πολλά κρατήματα δεν το πιστεύουν αυτό. Ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες δεν θεωρούνται αυτονόητες. Πολύ συχνά, ακόμα και σήμερα, στα κρατημέλη το στρατιωτικό προσωπικό θεωρείται ως άτομα τα οποία υπακούν, υπερασπίζονται αλλά δεν εκφράζονται. Μας υπερασπίζονται να εκφράζονται. Ακόμα και τα πρώτα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, οι κράτη που θεωρούν ότι οι ευρωπαϊκές αξίες είναι πολύ σημαντικές, ε, ακόμα και αυτά τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι το στρατιωτικό προσωπικό κάτι διαφορετικό, το βάζουν σε ένα άλλο επίπεδο τελείως χωριστά. Σε ειδικέ επιχειρήσεις, το είπα και στην αρχή, θα πρέπει να έχουμε κοινού κανονισμούς, ένα κοινό τρόπο για να αντιμετωπίζουμε το, τους στρατιώτες. Δεν συμβαίνει αυτό σήμερα. Μιλήσατε για τα εμβόλια, μιλήσατε για την ιατρική περίθαλψη, κατά τη διάρκεια της αποστολής, όταν μιλάμε για την ε, περίθαλψη, το θέμα μας αφορά πριν την αποστολή, κάτι τη αποστολή και μετά την αποστολή δεν αντιμετωπίζουμε, δεν δίνουμε την ίδια περίθαλψη σε όλου σήμερα. Ακόμα και αν πά στην ίδια αποστολή. Διαφορετικά άτομα από διαφορετικέ χώρε πάνε στην ίδια αποστολή, δεν έχουν ίδια περίθαλψη. Και θα πρέπει μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκείνου που μα υποστηρίζουν να υποστηρίξουμε ότι κάποια στιγμή, όταν στρατιώτε από διάφορε χώρε συμμετέχουν σε μία αποστολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν ένα ειδικό καθεστώ. Δεν μιλάμε για Ευρωπαίου στρατιώτε, γιατί ορισμένοι δεν έχουν όρεξη να ακούν αυτόν τον όρο, αλλά ως στρατιώτες που, που υπηρετούν, ε, που υπηρετούν την Ευρώπη και όχι μόνο τα κράτη-μέλη σε εκείνη τη φάση. Και μπορούμε λοιπόν με τη βοήθεια των εθνικών εμπειρογνωμόνων να προετοιμάσουμε αυτή την αποστολή από τη στιγμή δηλαδή, της προετοιμασίας να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή όσο χρόνο και αν πάρει. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε ανυπερθέτως και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κατάλληλο επίπεδο για να το κάνουμε. Το ΝΑΤΟ επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα. Σε επίπεδο ΝΑΤΟ κινείται περισσότερο προς τα κράτη-μέλη από ότι κινείται το ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα πιέζει τα κράτη-μέλη περισσότερο από ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην περίπτωση της Ισπανίας γνωρίζουμε το πρόβλημα το ισπανικό και τα προβλήματα σωρεύονται στις ένοπλες δυνάμεις της Ισπανίας. Το πρόβλημα των 45 ετών, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα στις ένοπλες δυνάμεις της Ισπανίας. Το συζητήσαμε το Ισπανικό Κοινοβούλιο και ελπίζω ότι η Ισπανία θα βρει μια λύση. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Δεν μπορεί κανείς να αφήνει εκτός κάποιους που υπηρέτησαν στι ένοπλε δυνάμεις, διότι κάποια στιγμή γίνονται 45 ετών. Δεν συμβαίνει μόνο στην Ισπανία, υπάρχουν και κάποιες άλλες χώρες που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Εμείς σαν EuroMill, δεν είμαστε κατά ε, των συμβολέων μικρής διαρκείας. Βλέποντας την αίθουσα, πιστεύω ότι το σύστημα που υπάρχει στη Γερμανία έχουμε στρατιώτε που υπηρετούν για κάποια έτη και μετά δημιουργείται ένα σύστημα, υπάρχει ένα σύστημα υποστήριξής τους. Θα υπάρχουν πάντα τέλειε. Δεν υπάρχει ένα σύστημα τέλειο. Υπάρχει σύστημα που υποστηρίζει τους στρατιώτες για να μπουν στην αγορά εργασίας μέσω κατάρτισης, υποστήριξης κλπ. Αλλά στις 45 να πούν τώρα τέλος, σας δίνουν 500 ευρώ το μήνα και για χαρά. Και ευχαριστώ πολύ, αυτό δεν είναι λύση δεν βοηθά τους ανθρώπους, δεν βοηθά τις αμυντικές δυνάμεις, διότι θα έχει σοβαρό πρόβλημα η Ισπανία να έχει επαρκές στατιωτικό προσωπικό. Αυτοί πρέπει να αποχωρήσουν, δεν θα αντικαθίσταται και αυτό επηρεάζει πολύ αρνητικά τη στατολόγηση προσωπικού της Ισπανικές Ένοπλες Δυνάμεις και εκεί πρέπει να συνεχιστεί η εποπτεία της καταστάσεως και χρειάζεται ευρωπαϊκή συζήτηση. Διερωτώ με πάντα γιατί για αυτά τα ζητήματα που είναι κοινά, αρκετά κοινά και συνήθισε αρκετές ενόπλες δυνάμεις στην Ευρώπη, γιατί να μην έχουμε μια τέτοια συζήτηση αυτού του τύπου, μαζί με το Ευρωκοινοβούλιο και τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Γνωρίζω ότι το κάνατε αυτό στο παρελθόν και κάποια δεδομένη στιγμή γνωρίζω ότι πολλά Εθνικά Κοινοβούλια δεν συμμετείχαν καν αλλά από την πλευρά σας, από πλευρά Ευρωκοινοβουλίου θα πρέπει να προσπαθήσετε να βρείτε έναν τρόπο ώστε τα εθνικά κοινοβούλια, εθνικοί βουλευτές να συμμετάσχουν σε αυτή τη συζήτηση και να μην γίνονται εθιμοτυπικέ επισκέψεις απλώ να συζητήσουμε τα κοινά προβλήματα και να βρεθεί ένας τρόπος προσεγγίσεω των προβλημάτων, κοινό τρόπο, πιο συντονισμένο τρόπο αντιμετώπιση. Η παρενόχληση, θρησκεία, πολύ γνωστά συστήματα για τις Ισπανικές Ένοπλες Δυνάμεις και όχι μόνο. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους που υπόκεινται σε σεξουαλική παρενόχληση. Παρακολουθούμε μια υπόθεση που αντιμετωπίζεται και εκτιμούμε την υποστήριξη από τα μέλη μας στην Ισπανία. Ναι, το άλλο είναι για τον συνάδελφο. Οι προσδοκίες που έχουμε μετά την υπόθεσή μας στην ε, Επιτροπή Κοινωνικής Χάρτας ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι περιπτώσεις είναι γνωστές. Έχουν συζητηθεί τα θέματα και με τα μέλη μας, διότι εκδικάζεται υπόθεση και εκδικάζεται μια υπόθεση μόνο όταν η κανονική συζήτηση και ο κοινωνικός διάλογος λείπει ή δεν δίνει αποτελέσματα. Στο τέλος προσφεύγει κάποιος στο δικαστήριο και δεν είναι η καλύτερη λύση. Αν είναι η μόνη λύση, τι να κάνουμε, αυτή είναι η λύση. Το να κερδίσει κανείς μία δίκη είναι ένα πράγμα. Μετά όμως, οι αλλαγές βάσει της δικαστικής αποφάσεων κάτι διαφορετικό. Το είδαμε στη Γαλλία. Στη Γαλλία, 2014, δύο υποθέσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το δικαίωμα ε, συνεταιρίζεστε στα, στο, στο προσωπικό των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων και ήξερε η Γαλλία ότι αν ε, υπέβαλε έφεση δεν θα κέρδιζε τη δίκη. Επέλεξε η Γαλλία να αλλάξει την νομοθεσία, να έχουν το δικαίωμα να συνεταιρίζεστε οι Γάλλοι στρατιώτε, οι Γάλλοι στρατιωτικοί. Αυτό είναι κάτι που ισχύει από το 2015 και αυτό που συμβαίνει είναι ότι από τα μέσα του 2015 το μόνο που άλλαξε είναι ότι έχουμε 11 συνδέσμους στη Γαλλία και κανείς δεν συμμετέχει στους συνεταιρισμούς αυτούς και ο μόνος λόγος είναι διότι δεν υπάρχει τίποτα πίσω από αυτό. Μπορεί να πεις σε μία ένωση και τελείωσε. Δεν υπάρχει κοινωνικό διάλογος. Δεν κρύβεται τίποτα, δεν υπάρχει κάποιο νόημα στη συμμετοχή. Γι' αυτό το θέσαμε επιτάπητο στο θέμα, το συζητούμε με τη Γαλλία οι ε, με τις στρατιωτικές ενώσεις στη Γαλλία που κατανόησαν ότι δεν πρέπει να ε, διχάζονται και να ενωθούν, να δημιουργήσουν μεγαλύτερες ομάδες για να μπορούν να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των στρατιωτικών. Το να κερδίσει μια δίκη, αυτό είναι κάτι. Αλλά μετά η υλοποίηση των αποτελεσμάτων που απορρέουν από την απόφαση κάτι άλλο. Έχουμε, περιμένουμε στην Επιτροπή Κοινωνικής Χάρτας να λυθεί το θέμα της Ιρλανδίας χρειάζεται ακόμα περισσότερη συζήτηση στην Ιρλανδία πριν να μπορέσουν οι σύνδεσμοί μας να μπορέσουν να πετύχουν αποτελέσματα για τη συνδικαλίζες στην Ιρλανδία. Συνεχίζονται οι προσπάθειες. Πρέπει να, πρέπει να έχουμε πραγματικό κοινωνικό διάλογο και να μην έχουμε τέτοιες δίκε. δίκες. Συνταξιδοτικό σύστημα μετά το σύνδρομο, το τραυματικό σύνδρομο, το συζητήσαμε είναι το ίδιο για αυτή την ε, περίπτωση το πρόβλημα. Πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερο συντονισμός, να συλλεχθούν δεδομένα, πληροφορίες, να ερευνηθούν αυτές οι υποθέσεις των, του μετατραυματικού συνδρόμου. Πρέπει να γίνει συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν μπορεί κάποια στιγμή να επιστρέφουν στατιώτες στα σπίτια τους, στη χώρα τους, να φυλάξουν την ευρωπαϊκή σημαία και μετά να ισχύει μόνο ε, να μένει μόνο η γαλλική-γερμανική σημαία στη στολή τους και να παραμένει το πρόβλημα σε επίπεδο 100 μελών. Αυτό πρέπει να επανέλθει σαν πρόβλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να συζητηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συνεργασία Ευρωπαϊκή Ενώσεω ΝΑΤΟ και αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί διότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των αποστολών Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των αποστολών ΝΑΤΟ, αλλά σε αποστολές Ευρωπαϊκής Ενώσεως όλες οι αποστολές μας δεν είναι πάντα εύκολες, δεν είναι απλώς περίπατος, ελοχεύουν πολύ σοβαροί κίνδυνοι για αυτές τις αποστολές και εκεί θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες. Ευχαριστώ κύριε Γιάκοπ. Ο Βίλιαμ. Νομίζω ότι ο Εμμάνιουελ είπε σχεδόν όσα ήθελα να πω. Θα είμαι σύντομος. Με ρώτησαν ε, ποιες είναι οι μεγαλύτερες διαφορές προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταξύ κρατών της Ένωσης. Πιστεύω όπως και εσείς ότι η διασφάλιση κοινή αντιμετώπισης κατά τη διάρκεια αποστολών ε, δεν θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Δηλαδή οι ίδιες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, τα ίδια κρεβάτια, τα ίδια περίθαλψη, οι ίδιοι γιατροί κλπ. Αλλά οι δομές, ε, οι συνοδευτικές της αποστολής είναι πιο προβληματικές. Για παράδειγμα, δικαιοδοσία σε περιπτώσεις αδικημάτων. Εδώ μπορεί να υπάρχουν διαφορές και σύστημα δικαιοσύνης. Σε κάποιες ε, χώρες είναι ένα πολύ κλειστό σύστημα στρατιωτικής δικαιοσύνης. Σε άλλες χώρες ένα καθαρά πολιτικό σύστημα, ένα σύστημα πολιτικών δικαστηρίων. Η εναρμόνιση λοιπόν θέλει ακόμη δουλειά. Αν λοιπόν δύο στρατιωτικοί στην ίδια αποστολή, από διαφορετική χώρα. Μία από τις οποίες έχει πολιτικά δικαστηρία και άλλη στρατοδικία, εάν διαπράξουν το ίδιο αδίκημα, πώς θα υπάρξει παρόμοια αντιμετώπιση. Τι προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μέσω ενός συστήματος, για παράδειγμα, ανεξάρτητης στρατιωτικής δικαιοσύνης. Επίσης, παλέμαχοι και το μετατραυματικό άγχος, η διαταραχή μετατραυματικού άγχους. Μετά δηλαδή την ε, ενεργόδράση Θα πρέπει να έχουν περαιτέρω ε, επιδόματα για παράδειγμα. Αυτό θα δημιουργούσε διάφορες κατηγορίες ε, αποστρατευθέντων. Για παράδειγμα θα μπορούσαμε από κάποια κράτη της Ένωσης οι αποστρατευμένοι να έχουν περισσότερα δικαιώματα και περισσότερα επιδόματα από, από άλλους αποστρατευθέντες από άλλες χώρες του ΝΑΤΟ που δεν ανήκουν στην Ένωση. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα. Αν έχει κανείς διαφορετικά δικαιώματα ενώ έχει συμμετάσχει στην ίδια αποστολή. Όποιο συμμετέχει σε βεβαίω διεθνεί αποστολέ στο εξωτερικό, πολλέ φορέ ούτω ή άλλω λαμβάνει περισσότερα. Περισσότερα επιδόματα, καλύτερη αμοιβή. Υπάρχουν λοιπόν ε, ορισμένα ωφέλη από την συμμετοχή σε αυτές τις αποστολές. Αλλά κατόπιν ε, μετά την αποστολή τι γίνεται, πόσο παροτείνονται αυτά τα επιδόματα, αυτά τα ωφέλη. Κατόπιν βεβαίως κατάρτιση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βεβαίως ισχύει, υπάρχει παντού αλλά με πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις. Σε, σε κάποια κράτη ενημερώνονται απλώς γενικά για την ε, ύπαρξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ενώ άλλοι κάνουν πολύ πιο ενεργά αυτή την κατάρτιση με ασκήσεις μετά, με παιχνίδια ρόλων. Υπάρχει λοιπόν ε, ένα ελάχιστο επίπεδο κατάρτισης. Το προσωπικό πρέπει να έχει συμμετάσχει σε τέτοιες καταρτήσεις. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο ασκείται αυτή η κατάρτιση είναι πολύ διαφορετική. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Και τους δυο σα και για τις παρουσιάσεις και για τις απαντήσεις που ήταν τόσο λεπτομεριακές. Το θέμα αυτό, όπως σωστά τονίσατε, δεν το συζητάμε πρώτη φορά ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σίγουρα δεν θα είναι και η τελευταία. Ιδιαίτερα λόγω ε, της αλλαγής ε, των σεναρίων για καταστάσεις ε, άμυνας στην Ένωση. Πολύ ενδιαφέρουσες λοιπόν οι παρεμβάσεις. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερος. Οπότε κλείνουμε την ακρόασή μας για το θέμα αυτό και κλείνουμε και την πρωινή μας συνεδρίαση. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν στις 2.30 για τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής διάταξής μας. Ευχαριστώ πολύ.